Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήρθατε στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Σύντομη συνεδρίαση μόνο σήμερα το απόγευμα, αλλά με πολύ σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Καλωσορίζω λοιπόν και όσους έχουν έρθει στην ώρα τους και ελπίζω σιγά σιγά να γεμίσει η αίθουσα. Είδατε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, τότε γίνεται δεκτή. Ανακοινώσει του Προέδρου δεν έχω να κάνω, εκτός βέβαια από τις γλώσσες ε, εστονικά, λετωνικά, μαλτέζικα, ξυλοβενικά, τα οποία δεν έχουν διερμηνία. Οι υπόλοιπε γλώσσες υπάρχουν. Μετά περνάμε στο 3. Προφορική ερώτηση για την αποφυγή φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Μια ερώτηση του Ζωά Φερέρα που δεν εγκρίθηκε την προηγούμενη φορά. Βεβαίως τώρα υπάρχει συνένεση για το κείμενο της προφορικής ερώτησης που θέλουμε να στείλουμε στην Ολομέλεια. Γι' αυτό ρωτάω υπάρχουν αντιρρήσεις ε, κατά του κείμενου αυτού που έχει διανεμηθεί. Ωραία λοιπόν, τότε εγκρίνεται και θα στείλουμε αυτό το ερώτημα στην Ολομέλεια. Για το τι έχει γίνει από την ανακοίνωση του 2009 και μετά. Ναι, Ζωά Φρέρα θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση έγινε με τρόπο κατακαιρματισμένο και αυτό ακριβώς μας οδήγησε και στο να υποχρεωθούμε να τροποποιήσουμε την ημερομηνία ε, συζήτησης ε, στην Ολομέλεια γιατί ξέ, θυμάστε ότι την πρώτη φορά που συζητήσαμε το θέμα στους συντονιστές είχαμε πει ότι θα περάσει το ζήτημα αυτό στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Εν πάση περιπτώσει όμως πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να καταβάλουν κάποια προσπάθεια και μακάρι να συμφωνήσετε όλοι σε αυτό έτσι ώστε τουλάχιστον ε, να μην ξεπεράσουμε και το Μάρτιο στην Ολομέλεια του Μαρτίου δηλαδή, να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Κάνω μια έκκληση λοιπόν να μην μετατεθεί ακόμα περισσότερο η συζήτηση. Το Μάρτιο να μας απασχολήσει στην Ολομέλεια. Έχω υπογράψει την επιστολή ήδη προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου πως θα θέλαμε να είναι στην ημερήσια διάταξη. Ελπίζω να χωρέσει στην ημερήσια διάταξη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ωραία. Περνάμε τώρα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση Λεπάζ για την τροποποίηση της οδηγίας του 2001 που αφορά την δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροπημένων οργανισμών στην επικράτειά τους. Ξέρουμε βεβαίω την νομοθετική πρόταση της Κομισιόν και είμαστε συνομοθέτες, άρα θα πρέπει και εμείς να σχηματίσουμε άποψη. Η Κορίν Λεπάζ έχει συντάξει μια έκθεση, οπότε θα της δώσω τον λόγο. Κορίν, παρουσίασε την έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την τιμή αλλά και το μεγάλο βάρος να σας παρουσιάσω μία έκθεση επί της πρότασης που μας έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γάμματα όμικρον στην επικράτηση. Ε, σύμφωνα με τι διατάξει και του Συμβουλίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω ότι εδώ δεν θα κάνουμε συζήτηση για του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, Πρέπει να είμαστε σαφείς εδώ. Δεν αφορά το θέμα αυτό η συζήτηση. Θα συζητήσουμε ένα ερώτημα το οποίο μα έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή αν είναι απαραίτητο ναι ή όχι να επιτρέψουμε στις ε, ε, χώρες μέλη να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά τους. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι ένα ε, δογματικό θέμα να τοποθετηθούμε δηλαδή υπέρ ή κατά των ε, ε, οργανισμών αυτών. Επίσης δεν πρόκειται να θέσουμε ένα αμφιβάλλο το γενικότερο θέμα αντιμετώπισης των γάμματα φόμικρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως να δώσουμε ενδεχομένως τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ολοκληρώσουν το σύστημα αξιολόγησης με κάποια δικά του στοιχεία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει το αίτημα αυτό, γιατί έχει κάνει το κείμενο αυτό. Υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος Μπαρόζο ήδη από την ας πούμε προεκλογική του εκστρατεία ε, είχε εκφράσει ε, την επιθυμία, την βούληση μάλλον να δώσει τη δυνατότητα αυτή στα κράτη-μέλη. Είναι γεγονός ότι πολλές χώρες απαγορεύουν την καλλιέργεια γαματαφόμικρο στην επικράτειά τους. Ε, επίσης, 7 χώρες έχουν υποβάλει ρήτρες προστασίας όσον αφορά την καλλιέργεια αυτή. Αλλά αυτές οι ρήτρες δεν έχουν επιτύχει. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινή γνώμη ε, αντιμετωπίζει, ε, ίσως λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης, ίσως λόγω έλλειψης γνώσεων, αντιμετωπίζει με μεγάλη καχυποψία την καλλιέργεια γάμματα φόμικρων. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο αφορά τον τρόπο εφαρμογής της ε, οδηγίας. Εάν είχε εφαρμοστεί σωστά η οδηγία 2001 κάθετος 1, ε, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε λόγος να απαντήσουμε στο ερώτημα το οποίο μας τίθεται. Δεν θα ετίθετο καν το ερώτημα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνων. Υπάρχει μεγάλη λοιπόν διαφωνία όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης. Πολλό δε μάλλον που το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος το Δεκέμβριο του 2008 ομόφωνα, και το υπογραμμίζω γιατί δεν συμβαίνει πολύ συχνά, ομόφωνα λοιπόν, στο τέλος της Γαλλικής Προεδρίας είχε ζητήσει από την ΕΦΣΑ μια σειρά μέτρων που θα αφορούσε και την διαχείριση της διευθέτησης των αντιθέτων γνώσεων, ε, απόψεων, ε, τη διευθέτηση με, ε, αντιτιθεμένων συμφερόντων. Ε, μια σειρά λοιπόν ερωτημάτων τα οποία στην ουσία δεν απαντήθηκαν. Αφετέρου, στο θέμα αυτό υπάρχει και η οικονομική διάσταση. Τα κράτη-μέλη ζήτησαν να εφαρμοστεί η οδηγία όσον αφορά τις ε, εκθέσεις αξιολόγησης των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων έτσι ώστε οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν, θα ήθελαν μάλλον να αναπτύξουν την χρήση γαματαφόμικρων να έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Όμως αυτού του είδους η έκθεση τελικά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δεν υπευλήθη ούτε στο Συμβούλιο ούτε βεβαίως και στο Κοινοβούλιο. Επομένως, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ε, θέμα την ε, δυνατότητα που θα έχουν τα κράτη να περιορίζουν να απαγορεύουν την καλλιέργεια γαματάφ όμικρον. Και εδώ ακριβώς μπαίνουμε ε, στο θέμα ε, στην ουσία του θέματος. Το άρθρο 26.3 αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται ε, ε, οργανισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην αγορά ή να υπάρξουν προβλήματα υγείας ή κοινωνικά λόγω της χρήσης γάμματα φόμικρων. Δεν υπάρχει όμως σαφής ορισμός. Δηλαδή στην ουσία έχουμε μια αρνητική δηλαδή, προσέγγιση. Δηλαδή λέμε ότι δεν θα πρέπει να έχει επίπτωση στην υγεία και το γενικό συμφέρον. Έχουμε τρει δυνατότητε. Η πρώτη είναι να απορρίψουμε το κείμενο. Απλά. Ξέρω ότι είναι η θέση που παίρνουν κάποιοι συνάδελφοι. Ορισμένοι θα ήθελαν να απορρίψουν ολοκληρωτικά το κείμενο γιατί θεωρούν ότι πρόκειται εδώ ε, για μία κατάφορη παραβίαση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και ότι επομένως δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ε, μία μορφή επανεθνικοποίησης η οποία βεβαίως έρχεται σε αντίθεση με την εσωτερική αγορά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτήν την άποψη γιατί ε, παραμένει ε, και η ε, ευρωπαϊκή αξιολόγηση και η ευρωπαϊκή προηγούμενη πρώτερη αδειοδότηση και επομένως δεν υπάρχει κανένα πρόσκομα στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και εμπορευμάτων. Δεύτερη θέση. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν καθόλου ένα κείμενο το οποίο θα έδινε την δυνατότητα επικύρωση τη δυνατότητα καλλιέργεια των γάμματα φόμικρων. Δεν νομίζω ότι και αυτή είναι αποδεκτή θέση, διότι το δίκαιο είναι αυτό που είναι. Αυτοί που θέλουν να καλλιεργήσουν γάμματα φόμικρων μπορούν να το κάνουν και επομένω μπορούν να έχουν και την αδειοδότηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επομένω δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον πρώτο ή τον δεύτερο δρόμο. Έχουμε μια άλλη δυνατότητα. Μπορούμε να επικυρώσουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια πρόταση η οποία βεβαίως ε, είναι θεάρεστη διότι λαμβάνει υπόψη ε, τις θέσεις πολλών κρατών μελών αλλά παρουσιάζει κατά την άποψή μου δύο προβλήματα. Πρώτον δεν λύνει με κανένα τρόπο την κακή εφαρμογή της οδηγίας 2001 ε, κάθετος 1 διότι δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα αυτό. Ε, και νομίζω ότι από νομικής απόψεως η πρόταση της Επιτροπής ε, είναι ε, ασφαλής και άλλωστε και οι απόψεις νομομαθών και στο Συμβούλιο αλλά και στο Κοινοβούλιο δεν είναι θετικές όσον αφορά την διατύπωση της ε, ε, Οδηγίας Επιτροπής. Δηλαδή δεν υπάρχει νομική ασφάλεια, δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τα κράτη-μέλη ε, όσον αφορά την ενδεχόμενη απειλή προς το γενικό συμφέρον. Νομίζω ότι εδώ αντιμετωπίζουμε λοιπόν μια πραγματική δυσκολία. Υπάρχει και μια τρίτη λύση, δηλαδή να τροποποιήσουμε την πρόταση της Επιτροπής και άλλωστε αυτή είναι και η πρόταση που σας υποβάλλω. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να εντάξουμε κάποιες απόψεις των κρατών μελών, έτσι όπως εκφράστηκαν από την ομόφωνη θέση του Συμβουλίου του 2008, με τρόπο όμως ώστε να υπάρχει νομική ασφάλεια όσον αφορά τα κριτήρια βάσει των οποίων κάποιες χώρες μέλη θα μπορούσαν να περιορίσουν την καλλιέργεια γάμματα στην επικράτειά τους. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά. Είναι αρκετά. και τα, ε, τα αίτια είναι είτε περιβαλλοντικά είτε ε, γεωργο-αγρο-περιβαλλοντικά. Ε, Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό. Το να θέλει κανείς να μην αμφισβητήσει την αξιολόγηση της ΕΦΣΑ, εντάξει, συμφωνώ. Όμως υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν ε, στο φάκελο και νομίζω ότι θα πρέπει να το πούμε, να τα αναφέρουμε αυτά. Πρώτον δηλαδή τι γίνεται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο με ειδικά οικοσυστήματα και ειδικές περιφε... γεωγραφικές περιφέρειες. Ε, υπάρχει στην οδηγία. Deuxièmement, la prise en compte de l'impact de l'OGM στην οδηγία 2001-18 ε, επίσης ε, δεν λαμβάνονται υπόψη οι τοπικοί κίνδυνη όσον αφορά ε, την αντοχή των διαφόρων μικροοργανισμών ή εντόμων. Τρίτον, η ε, η μη ύπαρξη αναφοράς σε ειδικών εθνικών οικοσυστημάτων γιατί γίνονται μελέτες οι οποίες όμως δεν αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή, αφορούν, έχουν γίνει κάποιες μελέτες ε, ενδεχομένως ακόμα και σε άλλη ήπειρο. Επίσης, Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ε, οι γεωπονικές ε, ε, ιδιότητες, οι ειδικέ γεωργικές πρακτικές και βεβαίως εδώ παραπέμπουμε και σε διάφορα κοινωνικά κριτήρια τα οποία ανεφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις της 2018 και που δεν εφαρμόζονται. Όλα τα στοιχεία αυτά υφίστανται και ε, στο ε, ε, άρθρο 192 ειδικά δίνεται η δυνατότητα να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία αυτά και επομένως θα πρέπει να έχουμε επομένως μια αντιμετώπιση η οποία δεν θα είναι εξ αντικειμένου αρνητική, δεν θα έχουμε μια αρνητική προσέγγιση αλλά μια θετική αντιμετώπιση αξιολόγηση της ενδεχόμενης χρήσης γάμματα φόμικρων στην επικράτεια της κάθε χώρας και επομένω, ε, εγώ θα ήθελα να τεθώ υπέρ των αναφορών του άρθρου 192 όσον αφορά το περιβάλλον και την ε, δημόσια υγεία και επομένω, νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε απλώ να κάνουμε πιο ασφαλή την όλη κατάσταση αφενό και αφετέρου να την διασυνδέσουμε με την ύπαρξη στοιχείων και δεδομένων τα οποία απαιτούν εδώ και δύο χρόνια περίπου, τρία χρόνια μάλλον, ε, οι χώρε. και που προβλέπονται στην οδηγία 2001 18. Νομίζω ότι ε, αυτό είναι απλό, είναι μια απλή προσέγγιση η οποία μπορεί να ε, διασυνδέσει και την, ε, τις ανάγκες των κρατών αλλά και τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ε, επιτρέπει στο να μην καθαιρεθεί όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει ήδη οικοδομηθεί. Επίσης θα δίνει ελεύθερη δυνατότητα επιλογής ε, στις ε, χώρες μέλη βάσει όμως και των περιβαλλοντικών μελημάτων ε, όλων των κρατών μελών. Αλλά θα δίνει ταυτόχρονα και την δυνατότητα να σεβαστούμε κάποιες συγκεκριμένες επιλογές είτε για ορισμένες καλλιέργειες είτε για ορισμένες γεωγραφικές περιφέρειες. Αυτό τα ήθελα να πω. Μπορούν να γίνουν βεβαίω παρατηρήσεις από όλους, αλλά ε, να πω και δύο λόγια σχετικά με την γνωμοδότηση τη Επιτροπής Γεωργίας για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι είναι Ενδιαφέρον, ενδιαφέρουσα η πρότασή τους να γίνουν, ε, ε, αυτό που προτείνει δηλαδή ο George Lyon, ε, να γίνουν υποχρεωτικές, υποχρεωτικοί κανόνες συνύπαρξης. Πιστεύω ότι γίνονται και κάποιες προτάσεις διαδικαστικά ορθές όσον αφορά την ασφάλεια του, του δικαίου. Απ' την άλλη πλευρά δεν ε, ε, συμφωνώ με το τρίτο σημείο όσον αφορά την ε, μόλυνση των σπορών γιατί νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον επικίνδυνο σαν βήμα. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε όσο πιο συνοπτικά μπορούσα και αυτό είναι το θέμα το οποίο το ζήτημα που σας υποβάλλω σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ Κορίν. Ευχαριστούμε για όλη αυτή τη δουλειά που έκανες και για την παρουσίασή σου. Το θέμα δεν είναι να δεχτούμε ή να απορρίψουμε, αλλά να δεχτούμε έναν θετικό κατάλογο με επιχειρήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη για να απορρίψουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Έτσι συνοψίζω την πρότασή σου. Έχουμε πάντα πρόβλημα με το χρόνο. Γιατί στις 4 πρέπει να έχουμε τελειώσει τη συζήτηση αυτή. Άρα τρία λεπτά έχουν οι σκιώδεις συζητητές, υπόλοιποι δύο λεπτά ο καθένας για τη συζήτηση. Λοιπόν, ποιος θέλει το λόγο. Πείτε το τώρα ή αλλιώς σιωπήστε για πάντα. Ποιος θα πάρει το λόγο. Θα διαβάσω τον κατάλογο. Κατρίν Σουλή, τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ενθαρρύνω την Κορίν Λαπάς γιατί πραγματικά ασχολείται με ένα δύσκολο θέμα γύρω από το οποίο γίνονται πολλές συζητήσεις. Την ευχαριστώ επίσης που μας ε, άκουσε όλους πολύ υπομονετικά. Το θέμα της επικουρικότητας είναι κάτι που στηρίζει τελικά μια εθνική αντιμετώπιση του θέματος και αυτό εμένα με ενοχλεί. Ως ευρωβουλευτές εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα, στέρεο, που να σέβεται βέβαια συγχρόνως τα κράτη-μέλη, τους αγρότες και τους καταναλωτές. Η επικουρικότητα είναι, όπως σας το να παραδεχόμαστε την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ότι μετά από την κρίση του ευρώ να επιστρέφουμε για αυτό το θέμα στην επικουρικότητα. Αυτό ήταν το πρώτο που είχα να πω. Το δεύτερο. Χρειάζονται πολύ στέρεα νομικά επιχειρήματα για να απαγορεύσουμε σε εθνικό επίπεδο την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Βλέπετε, μπορεί να υπάρξουν πολλέ και διάφορε διαμαρτυρίε και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην επιχειρηματολογία, να μην είναι υποκειμενική, να μην είναι αόριστη. Πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα επιχειρημάτων. Αυτό που προτείνει η Κορίν δεν νομίζω ότι μας προστατεύει από προσφυγές από κάθε πλευρά. Οι αγρότες μπορούν να τα βάλουν μαζί μας, όσοι ετοιμάζουν προϊόντα για τη βιοτεχνολογία κτλ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το θέμα των εισαγωγών. πώς θα μπορούσαμε να οικοδομήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα αν αφήνουμε απ' έξω ένα μέρος του προβλήματος που είναι ακριβώς εισαγωγές. Η σχετική τροπολογία θα έπρεπε να γράφεται γενικότερα στα πλαίσια της οδηγίας για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Συμφώνω πάντως με την Κορίν όταν αναφέρεται στο ισοδύναμο τι άλλο να προτείνουμε ανταυτού. Δεν λέω ότι έχω κάποια λύση θέτω και εγώ απλώς την προβληματική αυτή. Και το τελευταίο είναι λίγο πολύ αυτό που έλεγα και στην αρχή, ότι το κείμενο αυτό πρέπει να είναι απόλυτα συνεκτικό με την ε, κοινή γεωργική πολιτική και θέτει και το θέμα της ανταγωνιστικότητας των αγορωτών μας. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα ίδια ασφάλματα. Ξέρετε ότι στο Παρίσι είχαμε το σαλόνι της Γεωργίας, όπως το λέμε, μια έκθεση για την Γεωργία. Και εκεί οι αγρότες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την στρέβλωση του ανταγωνισμού. Μη λοιπόν μπούμε σε μια τέτοια κατάσταση και με τα γενετικά τροπημένα, τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς, όπως και γίνει με τα εντομοκτώνα. Παλέσκης τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια κάποια εμπειρία όσον αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Εδώ και αρκετά χρόνια μάλιστα. Και δεν συλλεύω καθόλου την Επιτροπή. Στη σημερινή κατάσταση η Επιτροπή καλείται να πάρει αποφάσεις παρόλο που δεν υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις. Με αυτήν εδώ την πρόταση και πάλι την ευθύνη τελικά την παίρνουν τα κράτη-μέλη. Με άλλα λόγια, αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα τα κράτη-μέλη. Είναι καλό αυτό? Τελικά κανένας δεν έχει να κερδίσει και ούτε περισσότερη νομική βεβαιότητα προσφέρουμε σε κανέναν. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να εξετάσει τελικά το θέμα από την στραβή οπτική γωνία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Κομισιόν θα έχει ικανοποιητικά επιχειρήματα. Τις αμφιβολίες αυτές τις έχουν θέσει και από την πλευρά της νομικής υπηρεσίας ε, του Κοινοβουλίου. Συνεπώς, είμαι υπέρ της θέσης της εισηγήτριας, δηλαδή να συμπεριλάβουμε τα θέματα του περιβάλλοντος σε έναν κατάλογο με επιχειρήματα υπέρ της απαγόρευσης. Και η κοινή γνώμη γνωρίζει περί γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και το δικό μας το σώμα το κοινοβούλιο βρίσκεται κοντά στον κόσμο και πρέπει να λάβει υπόψη του την κοινή γνώμη, τι θέλει και τι δεν θέλει. Να λάβουμε υπόψη μας τις ανησυχίες του κόσμου δηλαδή, συγχρόνως βέβαια να ενισχύσουμε την έρευνα, την σήμαση των προϊόντων και τα επιστημονικά δεδομένα. Κάθε χώρα που αποφασίζει υπέρ των γενετικά τροπευμένων οργανισμών πρέπει να παρουσιάζει μια αξιόπιστη στρατηγική που να λύνει τα προβλήματα επιμόλυνσης και να μας ε, διασφαλίζει καθαρά, καθαρές καλλιέργειες χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτό είναι πολύ βασικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μείνει ε, από την άλλη μία νησίδα απομονωμένη. Πολλοί επιστήμονες έχουν ήδη εκφραστεί και έχουν πει ότι πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τη χημία. Τι εννοούνε? εννοούν ότι είναι λιγότερο ευλαβεροί γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί από τα ντομοκτώνα. Να λοιπόν πώς περιπλέκεται το θέμα. Σίγουρα θέλω την κοινοτική προσέγγιση, αλλά σε αυτήν τη συγκεκριμένη κατάσταση που εξετάζουμε σήμερα, πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να βάλουμε σε αντίθεση ε, τα συμφέροντα και να τεθούμε αντίθετοι από τα συμφέροντα των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την κυρία Λεπάζ για την προσπάθειά της, για το γεγονός πως με τους σκιώδεις ηγητές συναντηθήκαμε δύο φορές στο Στρασβούργο και πληροφορηθήκαμε για τα σχέδιά της. Εξ ονόματος ομάδα δεν μπορώ να πω τίποτα ακόμα. Η κυρία Λεπάζη είπε πω ίσω καταθέσουν ακόμα κάποιες, ε, κα, καταθέσουν ακόμα ε, Το κοιτάμε αυτό. Δεν μπορούμε να... Δεν μπορώ να σα πω τι θα κάνουμε ακόμα ως προ αυτό. Σκεφτόμαστε και θα το δούμε το ζήτημα αυτό αργότερα στην εβδομάδα. Αλλά Θα ήθελα να πω το εξή. Εδώ πέρα συμφωνώ με την κυρία Λεπάς πως θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, πρόταση αυτή της ε, Κομισιού, θα πρέπει να έχουμε ένα καλό νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο μπορούν να συμβούν ε, όλα αυτά. Και βεβαίως είναι καλή η έκθεση. Βεβαίως η κρίσιμη τροπολογία είναι η 8 επί του άρθρου 28 που θα πρέπει βεβαίως να την ε, δούμε πιο λεπτομερώς. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε τα κριτήρια όσον αφορά το περιβάλλον, τα κριτήρια της υγείας επίσης, τα οποία θα τα προσπαθήσουμε να τα περάσουμε μέσω τρόπολογιών. Επίσης, κάποιες σκέψεις για το ότι τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνη και αρμοδιότητα για την προστασία της γεωργικής γης, ε, της χλωρίδας και της πανίδας και θεωρούμε πως ε, κάποιες ε, τροπολογίες θα πρέπει να καταθούν προς ενίσχυση του κειμένου της κυρίας ε, Λεπάς. Παραδείγματο χάρη για το ότι υπάρχει μία αβεβαιότητα όσον αφορά τον αντίκτυπο των περιβαλλοντικό ε, όσον αφορά το, τις δυνατότητες που δίνει αυτό το κείμενο. Παραδείγματος χάρη το ότι δεν υπάρχουν πλήρη δεδομένα για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των γενετικά τροπημένων οργανισμών στη χρήση των εδαφών, στη βιοπικιλότητα, στον πληθυσμό. Όλες αυτές θα είναι αρνητικές επιπτώσεις. Σκέφτομαι και ένα τρίτο κριτήριο το να προλάβουμε την ε, ανάπτυξη αντίστασης ε, στα εντομοκτώνα. Επίσης ε, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά βέβαια και να τα γράψουμε με μια νομική μορφή αλλά ένα κριτήριο θα μπορούσε να είναι παραδείγματος χάρη το να προλάβουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία από την ε, μη αηφόρο γεωργία. Επίσης ένα άλλο κριτήριο θα μπορούσε να είναι η προστασία γεωργικών πρακτικών που προωθούν την οικολογική αηφορία. Δηλαδή όλα αυτά είναι κάποιες προσεγγίσεις ε, στις οποίες θα μπορούσαμε να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες ε, για να ενισχυθεί η αρχική προσέγγιση της κυρίας Λεπάς και τα υπόλοιπα να τα σκεφτούμε ακόμα πολύ. Ευχαριστώ. Γιούρι μετά. Ε, ευχαριστώ για διαφορετικούς λόγους και εγώ δεν έχω κάποια θέση ιδιαίτερη της ομάδας μου. Κοιτάξαμε πολύ προσεκτικά την πρόταση. Συγχαίρω την Κορίν για τη δουλειά που έκανε, η οποία βεβαίως ήταν πάρα πολύ καλή και συμπεριέλαβε όλες τις απόψεις, αλλά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να πάει η σκέψη μας, πάντα φαίνεται πως υπάρχουν κάποιες ε, παρακάμψεις ή αδιέξοδα που μας οδηγούν ξανά στο συμπέρασμα πως η πρόταση αυτή δεν λύνει τίποτα αλλά μάλλον ε, ανοίγει και αποτελεί αιτία για ακόμη περισσότερες ε, διαφωνίες ε, και δεν μας δίνει αυτό το οποίο θέλουμε, αυτό το οποίο θέλουμε η Επιτροπή και ελπίζω και όλοι μας, δηλαδή ένα λογικό τρόπο για να προχωρήσουμε στην καλλιέργεια γενετικά τροπημένων οργανισμών στην Ευρώπη. Αν είναι να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, ανεξαρτήτως βεβαίως της δουλειά που έχει κάνει η Κορίν, δεν ξέρω το αν θα ακολουθεί τελικά αυτή η πορεία και εγώ είμαι διατεθειμένη βεβαίως να προσπαθήσω να καταθέσω τροπολογίες για να γίνει πληρέστερη αυτή η εργασία. Είναι σαφή αυτά τα οποία σας είπα, αλλά είμαι ειλικρινής και με ενδιαφέρον θα ακούσω και τους άλλους. Και εγώ οπωσδήποτε στην συνάντηση των ε, σκιωδών εισηγητών ε, και εγώ θα έλεγα πως θα έπρεπε να το απορρίψουμε ε, όλο το, κατασκεύασμα γιατί δεν μας δίνει κάποια νομική βεβαιότητα και έχοντας μεταβάλει αρκετέ φορές άποψη νομίζω πως εκεί καταλήγω ξανά. Thank you. Κάτι καλό τώρα. Ευχαριστώ. Θέλω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ ειλικρινά την κυρία Λεπάζ με το κείμενό της. Στην αρχή, όταν είδα την θέση της Επιτροπής, Πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω συζητήσει με την ομάδα μου ακόμα, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι η δουλειά που έκανε η συγγήτρια είναι πάρα πολύ καλή δουλειά. Θέτει πολύ σωστά τα ζητήματα. Οπότε πραγματικά συγχαρητήρια κυρία Λαπάζ από την ομάδα μας. Όταν είδα λοιπόν την πρόταση της Επιτροπής, είδα ότι έδινε περισσότερες αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη. Οπότε αυτό καθεαυτό αν τα κράτη-μέλη μπορούν να απαγορεύσουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο εδαφό του, θεώρησε ότι είναι καλό. Αλλά μετά είδα ότι τελικά η ευθύνη περνάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη. Και άρα και τα διάφορα προβλήματα ή οι δυσκολίες που ενδεχόμενα θα συναντήσουμε περνάνε από την Ευρώπη στα κράτη-μέλη και έτσι τελικά τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να κάνουν ε, τίποτα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εφόσον έχουν τα κράτη-μέλη την αρμοδιότητα, αυτό θα πρέπει να είναι μια πραγματική αρμοδιότητα, ώστε να μπορούν συνολικά να αναλάβουν την ευθύνη να απαγορεύσουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, οργανισμών στο έδαφό τους και να μπορούν και στη συνέχεια να διαχειριστούν την απαγόρευση αυτή. Έπειτα, ως αιτιολογία, πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη βάση επιχειρημάτων που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την υγεία. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το κείμενο. Έπειτα, το θέμα της εμπιστοσύνης του καταναλωτή είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 60% των Ευρωπαίων δεν νιώθουν καλά με την ιδέα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Οπότε αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεσή μας. Να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Μέχρι τώρα, σε αυτό το σημείο, το κείμενο της Επιτροπής είναι πολύ ασαφές, πολύ γενικό όσον αφορά την ε, ασφάλεια, ε, την υγεία και την θέληση των Ευρωπαίων καταναλωτών. Τέλος, πιστεύω ότι υπάρχουν και κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που τίθεται με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Στην ε, Ινδία, για παράδειγμα, Είδαμε τι γίνεται με τα δικαιώματα πατέντας και πόσο επηρεάζουν τη φτώχεια και την κατάσταση. Κάτι ακόμα έχω να πω, διακόπτει ο πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής. Ε, Κύριε Ρος, ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, βέβαια λυπούμαστε γιατί έχουμε πάντα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και δεν είναι σωστό όταν έχουμε τόσο σημαντικά θέματα. Εν πάση περιπτώσει μέσα στο μικρό χρόνο πρέπει να πω ότι το κείμενο αυτό ε, εάν παραμείνει όσοι έχει το κείμενο της Επιτροπής θα είμαστε απολύτως αντίθετοι. Εάν όμως καταφέρουμε να περάσουμε τις τροπολογίες ε, κατά την έννοια των προτάσεων της εισηγητρίας ε, θα είμαστε ευτυχείς. Θεωρούμε ότι η εισηγητρία έκανε εξαίρετη δουλειά. Κυρίως δε τη, η τροπολογία η οποία είναι η τροπολογία 5, η τροπολογία 4 σχετικά με το αρχείο το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί επίσης και αν περάσει και η τροπολογία 8, τότε σαφώς θα ε, υπερψηφίσουμε το κείμενο αυτό στην <coughs> Επιτροπή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Βλέπω πως ε, δεν θα το εξαντλήσουμε σήμερα. Γι' αυτό προτείνω να ακούσουμε την Κομισιόν μετά τους ομιλητές που έχουν λάβει το λόγο και τη Δευτέρα στο Στρασβούργο στην έκτακτη συνεδρίαση να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση για να δώσουμε την ευκαιρία και στου 7-8 ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο να μιλήσουν. Θα ακούσουμε λοιπόν τον ε, κύριο Μίκο, ο οποίο είναι αναπληρωτής διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Δράτω με τις ευκαιρίες να πω πως είναι η πρώτη μου συνεδρίαση υπό τη νέα μου ιδιότητα στην ε, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών. Όσον αφορά την πρόταση, πρέπει να επαναλάβω πως η πρόταση αυτή γράφτηκε από την Κομισιόν γιατί θέλουμε να αντικατοπτρίσουμε πιο ρεαλιστικά την ε, κατάσταση γιατί όπως είπατε υπάρχει ένα αδιέξοδο και αντικατοπτρίζουμε βέβαια τι απόψει των Ευρωπαίων πολιτών και κρατών μελών για να δώσω ήδη μια πρώτη απάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Λεπάζ για την έκθεση και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι δεν υπάρχει πρόταση ε, απόρριψης εδώ πέρα. Και θα ήθελα να πω πριν περάσουμε σε όλες τις ε, τροπολογίες ε, να αντιδράσω σε κάποιες από τις ιδέες που ακούστηκαν. Πρώτα απ' όλα το θέμα των υποχρεωτικών μέτρων συνύπαρξης που δεν ήταν στην πρόταση της Κομισιόν. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω από πού προέρχεται κάτι τέτοιο. Είναι παρόμοια θέση με αυτή την οποία είχε η θέση Γεωργίας, αλλά οπωσδήποτε είναι προς εξέταση από την Επιτροπή τα άλλα ζητήματα που αφορούν γενικώ τις ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχω κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα η πρόταση αυτή έγινε για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα τα οποία δεν υπάρχουν ήδη στην νομοθεσία και δεν έχουν αξιολογηθεί. Οπότε λέμε πως δεν θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε ξανά την σχέση με περιβαλλοντικούς κινδύνους ή κινδύνους για την υγεία. Γιατί το... υπάρχουν πλαίσιο μας δίνει κάθε επιλογή για να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε είναι διαθέσιμο για να δούμε στην αξιολόγηση κινδύνου ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την υγεία ή το περιβάλλον. Κάτι το οποίο, όπως είπε η κυρία Λεπάς, δεν θα αποτελέσει αντικείμενο της συζήτησης. Αυτό δεν σημαίνει, από την άλλη, πως δεν βλέπουμε άλλους πιθανούς λόγους που μπορούν να συνδέονται με το περιβάλλον και τους θεωρούμε εκτός πεδίου εφαρμογής. Προφανώς δεν είναι θετικός αυτός ο κατάλογος, είναι περισσότερο ενδικός όπως είπατε κυρία Λεπάζα, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να πω πώς έχουμε αυτό τον ενδεικτικό κατάλογο που ε, μας δείχνει τι εξετάζουμε εδώ πέρα, ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι και θα έλεγα πως ε, στο τέλος βεβαίω πάντα μπορούμε να συζητήσουμε, να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα είναι μέρος πρότασης, αλλά δεν νομίζω πως θα είμαστε σε θέση να καταρτήσουμε πλήρη κατάλογο όλων των πιθανών αιτίων, γιατί βεβαίως δεν μπορούμε να προβλέψουμε όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στην χύψη περιοχή κράτους μέλος. Συνοψίζοντας λοιπόν, εάν Σαφώς δεν υπάρχει σχέση και ζήτημα στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου. Ε, τότε είμαστε βεβαίως ε, στο πλαίσιο αυτής της πρότασης. Όσον αφορά την ε, απουσία αξιολόγησης, δεν το αντιλαμβάνουμε αυτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση χωρίς πληροφορίες κάναμε αποδεκτές αξιολογήσεις και δεν είχαμε τις ε, σχετικές πληροφορίες. Εάν υπάρχουν πληροφορίες που δεν υπάρχουν στο φάκελο, όπως είπαμε, το υπάρχον πλαίσιο επιτρέπει συνεισφορές ε, από ε, νέα επιστημονικά ή άλλα ερωτήματα. Εάν κάτι προέκυψε μετά από την διαδικασία, υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι ρήτρε διασφάλισης, οι οποίες υπάρχουν ήδη. Δεν βλέπουμε κάποιο λόγο να αλλάξει η πρόταση. Από την άλλη, η τρίτη ομάδα επιχειρημάτων για τη χρήση γης, χωροταξία κτλ. Όλα αυτά πηγαίνουν πάρα πολύ κοντά στις προτάσεις μας σε σχέση με την ενδεικτική λίστα, οπότε είμαστε πάρα πολύ δεκτικοί στο να βρούμε μια κατάλληλη διατύπωση εδώ πέρα. Επίσης υπάρχουν κάποια πράγματα στην πρότασή σας ε, που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις και αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν πολλά ζητήματα που σχετίζονται με τους γενικά τροπημένους οργανισμούς όπως η συνύπαρξη, αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων. Να σας πενθυμίσω εδώ πέρα πως ε, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές ε, συντάσσονται αυτή τη στιγμή. Προφανώς μπορείτε κι εσείς να λάβετε μέρος στη διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω γιατί πρέπει να αναφερθεί σε αυτήν εδώ πέρα την πρόταση. Ευχαριστώ. Να ευχαριστούμε κύριε Μίκο και καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας ε, στην πρώτη σας εμφάνιση με ένα μεγάλο θέμα Λοιπόν, η ότι Ρότμπερντ έχει συνεδρίαση του Προεδρείου μετά, οπότε νομίζω καλό είναι να την ακούσουμε τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αν και παραδέχομαι πως ε, θα ήθελα να παρακολουθήσω ολόκληρη τη συζήτηση. Μετά από αυτά τα οποία είπε η κυρία Λεπάζ, θα ήθελα να αναφέρω δύο συγκεκριμένα σημεία. Εάν αλλάξουμε κάτι στην οδηγία περί απελευθέρωσης, δηλαδή αν πρέπει να υπάρξει ρητή αδειοδότηση ενός προϊόντος, ε, η οποία μπορεί πλέον από κάποιες χώρες να αξιολογηθεί διαφορετικά ή να μην την λάβουν υπόψη κάποιες χώρες, τότε αυτό έχει νόημα μόνο εάν κάτι τέτοιο όσον αφορά τους λόγους υγείως η περιβάλλοντος αφορά συγκεκριμένα το κράτος μέλος. Αλλιώς μιλάμε για ανταγωνισμό της ΕΦΣΑ, γιατί η ΕΦΣΑ κάνει μια αξιολόγηση, με βάση αυτό δίνει την άδεια η Κομισιόν και αν δεν λαμβάνει μέρος σε αυτό μιας, μια, ένα κράτος μέλος, είναι δικαίωμά του. Αλλιώς θα καταλήξουμε σε έναν ανταγωνισμό τον οποίο δεν θα κερδίσει κανένα κράτος μέλος. Δεύτερον, το οποίο, επειδή πιέζει και ο χρόνο, είναι βέβαια το ζήτημα τη επιμόλυνση. Η κυρία Λεπάζη είπε πω ε, θεωρεί πω πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λόγω των οικονομικών προβλημάτων για του γεωργού. Εγώ έχω κάπως διαφορετική άποψη γιατί ξέρετε πως ε, δώσαμε αγώνα για το όριο επιμόλυνσης με τα Novel Foods. σε μια πυκνοκατοικημένη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τελείως διαφορετικές απόψεις τα κράτη-μέλη υπάρχουν μόνο δύο δυνατότητες. Πρώτον, ένας κανονισμός συνύπαρξης και απόστασης που πρέπει να είναι δεσμευτικός και εδώ πέρα η Κομισιόν λάθος έκανε και δεν το έφερε εδώ πέρα μέσα στην πρότασή της. Πρέπει να υπάρχει, δηλαδή όσοι δίνουν την άδεια θα πρέπει να τηρούν αν έχουν μια γειτονική χώρα η οποία δεν θέλει να τα αφήσει τους γενετικούς τροπημένους οργανισμούς, να τηρούν κάποιους περιορισμούς. και νομίζω έτσι θα, θα μπορέσει να ε, ε, ασκήσουμε και την ε, απαραίτητη πίεση. Αυτά και τελειώνω εδώ πέρα γιατί ξέρετε θα μπορούσα να μιλήσω ακόμη πέντε λεπτά. Ο πρόεδρος. Ναι βεβαίως ε, μιλήστε δύο λεπτά και θα έχετε άλλα τρία λεπτά στις τροπολογίες. Ο Ρίχαρτ Ζέμπερ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Καλωσορίζω την πρόταση της Κορίν Λεπάζη ιδιαίτερα γιατί Βλέπετε πως υπάρχει μεγάλη επιστημονική αβεβαιότητα όσον αφορά αυτή την οδηγία και νομίζω πως η άποψη της ΕΦΣΑ δεν είναι κάτι το θέσφατο. Υπάρχουν ε, άλλες απόψεις οι οποίες δεν υπάρχουν μέσα σε αυτή την ε, αξιολόγηση. Υπάρχουν λοιπόν και κάποια περιφερειακά στοιχεία τα οποία ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αλλά νομίζω πως θα πρέπει και υπάρχουν επιστημονικοί λόγοι να δώσουν περισσότερες δυνατότητες στα κράτη-μέλη να περιορίσουν την καλλιέργεια. Το δεύτερο και αφορά βεβαίως τις ανησυχίες των ε, πολιτών ε, και ακούμε πως 60% των συμπολιτών μας είναι κατά, νομίζω πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Οπότε θεωρώ πως σωστό θα ήταν, όπως είπε και η κυρία Λεπάζ, να επεκτείνουμε αυτούς τους επιστημονικούς λόγους και στην πτυχή της υγείας και του περιβάλλοντος και να δώσουμε περισσότερα δικαιώματα στα κράτη-μέλη. Νομίζω πως είναι πολύ ρεαλιστική αυτή η προσέγγιση της ε, Κομισιόν, αν και σε κάποια σημεία χρειάζεται βελτίωση. Αλλά νομίζω πως πολιτικά αποτελεί απάντηση στο ερώτημα το πώς θα βγούμε από αυτή την κατάσταση, γιατί είναι ουτοπικό να πιστεύουμε πως ε, μπορεί κάποιος να εξαναγκάσει ένα κράτος μέλος, να καλλιεργήσει τέτοιους οργανισμούς. Και βεβαίως ε, θα γίνει ε, σιγά σιγά μεγαλύτερη και η αποδοχή του πληθυσμού, αλλά βλέπετε πως υπάρχουν εδώ πέρα μεγάλες συμφέροντα των εταιριών που θέλουν να προωθήσουν αυτά τα προϊόντα, οπότε πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα πως αυτό το ζήτημα είναι ζήτημα επικουρικότητας και υποστηρίζω εδώ πέρα την κυρία Λεπάζ. Ευχαριστώ. Ο Βιτόριο Πρόντι είναι μέλος και της ΣΤΟΑ και έχει να μας πει κάτι. Παρακαλώ. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ήθελα απλά να πληροφορήσω την Επιτροπή μας ότι σύμφωνα με την εντολή που μου είχε αναθέσει ως ε, μέλος εκπροσωπών ε, το, την Επιτροπή μας ε, στο ΣΤΟΑ, παρουσίασα το πρόβλημα, δηλαδή ότι μία μείωση ή περιορισμός της βιοπικιλότητας μπορεί να εκθέσει την ε, ανθρωπότητα στον κίνδυνο μείωσης της ποσότητας ε, ε, τροφής γιατί τα έντομα ή οι μολύνσεις μπορεί περαιτέρω να επηρεάσουν κάποιες ποικιλίε. Και βεβαίως όσο, περισσότερες, ε, όσο περισσότερο οι ποικιλίε αυτές στέφονται από επιτυχία όσον αφορά την απόδοση, τόσο μικρότερη ε, είναι η διοπικιλότητα και επομένως ο ευάλωτος χαρακτήρας ε, που θα έχουν πλέον αυτές οι ποικιλίε απέναντι στις μεταλλάξεις των μολύνσεων. Το θέμα αυτό θα απασχολήσει το ΣΤΟ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ. Vielen Dank, äh, Karl Schlüter. Ευχαριστώ, Καλ Σλίτερ. Νομίζω ότι πάει στη τη σωστή κατεύθυνση η Κορίν Λαπάζ. Έχω μια ερώτηση για την Επιτροπή, γιατί εγώ βρίσκω ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Η πρόταση σήμερα είναι ότι προκειμένου να το ξέρει το γενετικά τροποποιημένο οργανισμό η Κομισιόν θα πρέπει πολύ γρήγορα με πολύ σύντομες δοκιμές οι αρμόδιοι να αποδείξουν ότι είναι επικίνδυνος αυτός ο γενετικά τροπευμένος οργανισμός ε, για τον κόσμο. Και ότι πρέπει μια αρνητική γνωμοδότηση να δώσει και που δεν πρόκειται να δώσει ποτέ. Με, με ένα τόσο, μια τόσο μικρή δοκιμή δεν φτάνει. Έτσι κι αλλιώς δεν συνάδει όποιος γενικά δεδομένος οργανισμός με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής υπέρ ε, του κοινού, της βιοπικιλότητας κλπ. κλπ, Όμως ποτέ δεν έχει χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανένα άλλο κριτήριο πέρα από την ΕΦΣΑ. Πρέπει να το κάνει όμως, γιατί πρέπει να λάβει υπόψη της και την υπόλοιπη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τώρα 17 περιπτώσεις εκκρεμότητα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα κάνει θα πει ναι για τα όλα, θα αναλάβει τις ευθύνες της ποτέ. Θέλω να ξέρω τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Και η δεύτερη ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η εξή. Γιατί τα κράτη-μέλη πρέπει να ανακοινώνουν ένα μήνα πριν την απόφασή τους όλα τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή. Εντάξει, καλή διαφάνεια, αλλά γιατί τώρα. Γιατί, γιατί δεν θα έχει καιρό η βιομηχανία να κάνει το λόμπι της. Γιατί, γιατί τώρα. Και έπειτα γιατί έχουμε εδώ πέρα ένα άρθρο για τη δημοκρατία. Όπως απαγορεύουν πολλές χώρες ε, τα πυρηνικά, γιατί να μην κάνουμε το ίδιο και εδώ. Αν δημοκρατικά έχει ληφθεί απόφαση να μην χρησιμοποιούνται οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί σε μια χώρα, γιατί να μην μπορεί αυτή η χώρα να το αποφασίσει από μόνη της και χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Θα σταματήσουμε εδώ πέρα τη συζήτηση για την έκθεση της Κορίν Λεπάζ για τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς και θα συνεχιστεί Δευτέρα στο Στρασβούργο. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι στον κατάλογο και η Κορίν Λεπάζος, η εισηγήτρια βεβαίως, η οποία, θα, η οποία θα απαντήσει. Προθεσμία για τις τροπολογίες λογικά είναι μία μέρα αργότερα, στις 8 και όχι στις 7 Μαρτίου. 8 Μαρτίου μεσημέρι και Δευτέρα 7 και 15 στο Στρασβούργο είναι η δική μας συνεδρίαση για τα benchmarks και θα συνεχιστεί η συζήτηση για τους γενετικά προηγουμένους οργανισμούς. Λοιπόν, συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερής διάταξης. Ακρόαση για το θέμα μείωση των κλιματικών αερίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 20% και παραπάνω.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 So, liebe Kolleginnen Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήλθατε στην ακρόαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για το θέμα 20% και παραπάνω. Μείωση των ε, ριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020. Σημαντικό θέμα από αυτά τα οποία μας απασχολούν στην πολιτική, στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του κλίματος υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη συζήτηση αυτή και καλωσορίζω βεβαίω την κυρία Επίτροπο, την κυρία Χέντεγκαρτ. Καλώ ήρθατε, γνωστή στην Επιτροπή μας. Οι συγητές είναι Βεβαίω Μπας Άϊχουτ και η Ρωμάνα Ιωδαμψή σε λίγες με Επιτροπή Βιομηχανίας. Μετά βεβαίως καλώς και την Κομισιό και υπάρχει και η Ουγγρική Προεδρία και θα καλωσορίσω και τους ειδικού μας στους οποίους προσκαλέσαμε να μας δώσουν πληροφορίες για αυτό το επίμαχο θέμα ποια είναι τα ωφέλη, ποιο είναι το κόστος τι μπορεί να επιτευχθεί θα έχουμε τις επόμενες δύο μισή ώρες ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το θέμα. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε μέχρι το 2050. Αυτό το αποφάσισε βεβαίως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. με 95% μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Και ρωτιέται κανείς βεβαίως το αν και τι, πώς θα φτάσουμε σε αυτά τα υψηλά ποσοστά το 2050 η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την Κομεχάγη είχε προσφέρει ένα 30% εάν και άλλες χώρες ε, συγκρίσιμες έκαναν κάτι παρόμοιο. Το ερώτημα είναι αν αυτή η στρατηγική εξακολουθεί να ισχύει ή χρειαζόμαστε μια στρατηγική διαφορετική ε, για τον ένα ή τον άλλο λόγο ορίζω λοιπόν και θα δώσω τον λόγο στον Μπας Άικχουτ γιατί ξέρουμε όλοι το πιεσμένο πρόγραμμα και ζητώ συγγνώμη μετά θα αφαιρώ τον λόγο και τώρα θα δώσω τον λόγο στον Μπας Άικχουτ για να κάνει εισαγωγή 5 λεπτών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω λιγότερο από πέντε λεπτά. Γιατί σήμερα το απόγευμα το χρόνο μας πρέπει να το δώσουμε στους εμπειρογνώμονες που έρχονται από το χώρο της επιστήμης και που θα μας πούν πώς το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών μπορούν να βοηθήσουν, ποια είναι υπέρ, ποια είναι τα κατά, στον τομέα της υγείας και αλλού. Και να δούμε και τι γίνεται και σε διεθνές πλαίσιο. Οπότε, για του εμπειρογνώμονε είναι ο χρόνο μα σήμερα και εμεί οι Ευρωβουλευτέ είμαστε εδώ για να του ακούσουμε, να μάθουμε από αυτού και να του ρωτήσουμε πράγματα έτσι ώστε να πάρουμε όλε τι πληροφορίε που έχουν αυτή στη διάθεσή του. Όπω είπατε και εσεί, Πρόεδρε, Έχουμε θέσει μακροπρόθεσμους στόχους και εγώ θα προσθέσω εδώ και κάτι άλλο. Τους δύο βαθμούς στόχο. Ένας πολύ σημαντικός στόχος πάνω στον οποίο έχουμε συμφωνήσει ως Ευρώπη αλλά και στο Κανκούν σε διεθνές επίπεδο. Συμφωνούμε λοιπόν για το στόχο των δύο βαθμών και εφόσον συμφωνούμε γι' αυτόν θα υπάρχουν επιπτώσεις. Δηλαδή πρέπει να δούμε πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές μας. Η επιστήμη θα πρέπει να μας βοηθήσει. 80 με 90% λέμε για τις βιομηχανικές χώρες μέχρι το 2050 και 25 με 40 το 2020 για τις βιομηχανοποιημένες χώρες. Αυτό σημαίνει 50% ότι έχουμε πιθανότητες να πετύχουμε το στόχο των δύο βαθμών. Ακόμα δηλαδή και αν προχωρήσουμε με τη στρατηγική μας για να πετύχουμε το στόχο μας, μόνο 50% πιθανότητες έχουμε να τον πετύχουμε. Καταλαβαίνετε ότι το σκηνικό είναι ξεκάθαρο. Πολύ θα ήθελα να ακούσω, εννοείται και από την Εκοφής να μας πει πώς βλέπει την κατανομή του βάρους. Από την άλλη, τι σημαίνει για την οικονομία μας. Είμαι από τους πράσινους και Καταλαβαίνετε ότι με ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος, αλλά ακόμα και αν το δει από το οικονομικό πρίσμα, έχει νόημα να θέλουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Αν δούμε τις αγωγές πετρελαίου στην Ευρώπη, η σημερινή συζήτηση δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν στη Βόρεια Αφρική, αν προχωρήσουμε από το 20% στο 30% μείωση. Αυτό σημαίνει λιγότερες εισαγωγές πετρελαίου αξίας 40 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν μιλάμε 88 δολάρια το βαρέλι, παρόλο που ξέρουμε ότι σήμερα είναι πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Σημαίνει λοιπόν λιγότερες εισαγωγές πετρελαίου, άρα ε, μεγάλο οικονομικό κέρδος. Και για την υγεία το κέρδος θα είναι μεγάλο. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα τα δεδομένα από μένα, αλλά θα μπορέσουμε να μειώσουμε από 6 σε 35 εκατομμύρια ευρώ ε, το κόστος για την υγεία που δαπανάμε σήμερα. Θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε τι σημαίνει για τη βιομηχανία η αλλαγή αυτή του στόχου, τι σημαίνει για τις διάφορες χώρες. Αλλά θέλω να μας προτείνετε και λύσεις. Αν το κάνουμε αυτό και πάμε πέρα από το 20%, τι σημαίνει για το Ταμείο Συνοχής, τι σημαίνει για τις διάφορες χώρες και τι διορθώσεις μπορούμε να κάνουμε ώστε ε, στον τομέα του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών τι επιπτώσεις θα υπάρχουν. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Εμείς οι ευρωβουλευτές, όπως είπα και πριν, πρέπει να καθίσουμε να ακούσουμε και να κάνουμε ερωτήσεις. Εγώ αυτό θα κάνω. Η έκθεση θα δημοσιευθεί αυτή τη βδομάδα, μετά θα περάσουμε σε τροπολογίες και ελπίζω ότι τον Ιούνιο θα έχουμε μια ιδιαίτερη ισχυρή θέση ως Κοινοβούλιο για να περάσουμε τη συζήτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω, έχω κερδίσει ένα λεπτό, έχω μιλήσει ένα λεπτό λιγότερο. Ε. Περιμένω τη συνέχεια. Πρόεδρος, ναι, πράγματι, ευχαριστούμε που μας δώσατε ένα λεπτό. Η κυρία Γιόρνταν είναι εδώ από την ε, Σλοβενία. Αλλά πρώτα θα μιλήσει η Επίτροπος, η κυρία Κόνη Χέντεγκαρτ. Επίτροπος για θέματα δράση για το κλίμα. Για πείτε μας και εσείς τι ιδέες έχετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε για αυτήν την ε, ε, πρωτοβουλία που πήρατε σε τόσο όσο στη χρονική στιγμή. Γιατί είχαμε ε, το Σύμβουλο προηγουμένως το οποίο κατέληξε σε πολύ σαφή συμπεράσματα. Αναφέρεται σαφώς ότι έχει μειωθεί το κόστος της επίτευξης των ε, στόχων, τουλάχιστον σε αναθεωρημένη βάση ε, σχετικά με το 2008. Ε, το προηγούμενο Μάιο είχαμε μια ανακοίνωση σχετικά, αλλά από τότε είχαμε πολλές εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα τη θετική έκβαση της Κανκούν. Ξέρουμε ότι περισσότερες από 80 χώρες έχουν θέσει εσωτερικούς εγχώριους στόχους και αυτή τη στιγμή τότε Κομπεχάγης πλέον έχουν ενταχθεί ε, στην θέση και των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης και επίσης σαν ένα πρώτο συγκεκριμένο στόχο, αποτέλεσμα μάλλον σας λέμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει ο δικός χάρτης για το 2050 όσον αφορά τις εκπομπές. Βεβαίως λέμε ότι 80 μέχρι 95% θα είναι ο στόχος μείωσης των ρήπων και είναι σαφές και το λέμε ότι αν θέλουμε να έχουμε μια ε, σωστή οικονομική ας πούμε αντιμετώπιση θα πρέπει ε, το 80 95% να παραμείνει αλλά βεβαίως σε, σε εγχώριους στόχους ε, να έχουμε το τουλάχιστον 80%. Δεν είναι σοφό από άποψη οικονομική να συμφωνήσει κανείς ότι χρειάζεται μια μακροχρόνια ε, μεταβατική περίοδο στην οποία ε, θα ε, διοχετεύονται τελικά εκατομμύρια εκατομμυρίων στους κύριους ανταγωνιστές και επομένως είναι πιο οικονομικά σοφό να ξεκινήσει κανείς με αναέτος προγράμματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι ε, ε, θα πρέπει να βασιστούμε σε πρότυπα, στο modeling, το οποίο ε, θα πρέπει να γίνεται αναέτος. Έτσι ώστε όχι να έχουμε μονάχα το 80% μέχρι το 2050 σε χώριο επίπεδο, αλλά 40% μέχρι το 2030 και αυτό καταδεικνύεται σαφώς μέσα από τις μελέτες επιπτώσεων ότι μπορεί να γίνει και σε συνεργασία βεβαίως με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών και ε, για το 2020 20% μείωση ε, δεν είναι το περισσότερο που μπορούμε να κάνουμε. Ε, βάσει της άσκησης modeling ε, καταδεικνύεται ότι μπορούμε να φτάσουμε στο 25%. Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Μιλούσαμε προηγουμένως για τα εργαλεία Ε, μπορούμε λοιπόν να έχουμε μείωση 20% για το 2020, ε, μπορούμε όμως ε, να επιτύχουμε και το 20% για, τους, ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν έχουμε το 20% όσον αφορά την ε, τον στόχο ε, ενεργειακής αυτάρχειας. Εάν καταφέρουμε και το στόχο αυτό και εάν ε, διατηρήσουμε και όλους τους στόχους και τα σχέδια, τα προγράμματα που έχουν οι χώρες, τότε θα φτάσουμε άμεσα και χωρίς περαιτέρω προσπάθεια στο 25% της μείωσης. Με άλλα λόγια, δεν είναι τυχαίο ε, το ότι την επόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα κάνει ταυτόχρονα ε, και το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα αλλά και το σχέδιο για την, το χάρτη για την μείωση της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος. Πιστεύουμε απλώς ότι θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνει ο κάθε τομέας, δηλαδή που θα πρέπει να βρίσκεται ας πούμε η γεωργία για το 2015, 2020-2025, τι θα γίνεται με τη γεωργία, τι θα γίνεται με, την, ε, με τις μεταφορές, με τη βιομηχανία κλπ. λοιπά με όλους τους τομείς, δηλαδή τι θα πρέπει να προωθήσουν και πού θα πρέπει να φτάσουν οι διάφοροι τομείς, έτσι ώστε το 2050 να έχουμε επιτύχει τους στόχους μας. Πολλά εργαλεία ε, αναφέρονται, ας πούμε η τυποποίηση που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, εργαλείο Αναφέρονται και άλλα στην οδηγία. Επίση, ε, χρειαζόμαστε τιμολογική πολιτική έτσι ώστε τα κίνητρα να είναι σωστά και όπως ε, ε, επανειλημμένα καταδεικνύουν όλες οι μελέτες είναι ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία τακτική κύρωση των κακών και επιβράβευση των καλών. Το μήνυμα λοιπόν είναι σαφές. Ε, θα πρέπει να ε, ε, φορολογείται ακριβότερα αυτό που κες, να φορολογείται φτηνότερα αυτό που κερδίζεις. Tax more what you burn, tax less what you earn. Η καινοτομία επίση είναι σημαντικό θέμα. Έχει ήδη προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, την, ε, έχει προτείνει λέγω από πέρσι τη δημιουργία μιας ε, επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με τι διαφορέ ανάμεσα στο 13 και στο 20. Δεν σημαίνει ότι θα, υπάρχει, θα, θα προβλέψουμε ελεύθερη αδειοδότηση, αλλά ότι θα υπάρχει μια καλύτερη τιμολογιακή πολιτική και επομένως και στη, οι τιμέ των πληστηρισμών θα είναι καλύτερε. Το θέμα αυτό θα ήθελα να το θίξω εδώ εάν ασχοληθούμε μονάχα με την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα αλλά όχι με το θέμα του αριθμού αδειοδοτήσεων τότε ε, δεν θα έχουμε αντιμετωπίσει συνολικά το θέμα. Ξέρει πάρα πολύ καλά η βιομηχανία πώς μπορεί να γίνει πιο ελκυστική η όλη διαδικασία. Ε, στις επόμενες ε, ε, δημοσιονομικές προοπτικές επίσης θα πρέπει, και το έχω ξαναπεί άλλωστε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο το θέμα. Θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστική η ενεργειακή αποτελεσματικότητα για τις χώρες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το δυναμικό της γεωργίας γιατί πολλά μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Ένα τελευταίο πράγμα το οποίο ήδη αναφέρθηκε σε σχέση με την ε, βιομηχανία. Πέρσι ας πούμε εισαγάγαμε 70 ε, δις δολάρια επιπλέον αξία πετρελαίου από ό,τι την προηγούμενη χρονιά ε, και ε, πληρώσαμε ακριβότερα 14 δολάρια αναβαρέλι. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν βεβαίως ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όλο και λιγότερη ενέργεια τέτοιου είδους έτσι ώστε να οδηγηθούμε σιγά σιγά σε μια κοινωνία με χαμηλότερο διοξίδιο του άνθρακα. Και βεβαίω είναι σαφές ότι η φτηνότερη ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν καταναλώνει κανεί, η ενέργεια που δεν ε, χρησιμοποιεί ε, και ξέρουμε ότι υπάρχει αυξητική τάση τη τιμή ε, αυτού της μορφή ενέργειας, όχι γιατί συμβαίνουν αυτά στη Βόρεια Αφρική, αλλά γενικότερα είναι η τάση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Το μήνυμα είναι σαφέ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία ε, στον ε, κύριο Πίτερ ο Λέιχος. Uh, την κυρία Γιορμπάνη, η οποία αντικαθιστεί τον κύριο Λάχος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση από την πλευρά της Προεδρίας και εμείς θεωρούμε πως ε, αυτή η συζήτηση είναι κάτι το βασικό για την Προεδρία μας. Αλλά Βεβαίως γνωρίζουμε πως κάποια κράτη-μέλη ακόμα ε, δεν δέχονται το ότι πρέπει να δεχτούν ε, ένα νέο στόχο. Και βεβαίως αυτό σχετίζεται με την ε, τρέχουσα οικονομική κρίση και την πίεση που ασκεί στα κράτη-μέλη. Οπότε ως ε, Προεδρία πρέπει εμείς να διατηρήσουμε αυτές τις φιλοδοξίες. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρχει ευκαιρία για τα κράτη-μέλη να γίνει μια ενημερωμένη συζήτηση και να τους δώσουμε τις πληροφορίες που έρχονται από την Κομισιόν και πάω από παραέξω στις διεθνείς εξελίξεις όπως την έκθεση του είναι για την πράσινη οικονομία και την αναλογική έκθεση του ΩΣΑ. Θα δουν τα κράτη-μέλη λοιπόν πως δεν μιλάμε μόνο για εκπομπές αλλά και για την οικονομία και για το να επιτύχουμε τους στόχους του 2020. για να έχουμε μια Ευρώπη με καλύτερη χρήση πόρων. Για να το επιτύχουμε αυτό, το σχέδιο το οποίο είχε εγκριθεί ήδη στο Συμβούλιο του... θα εγκριθεί στο Συμβουλίο του Μαρτίου και βεβαίως αναμένουμε απάντηση του κυρίου Στάινερ ε, για το εάν θα έρθει να κάνει μία παρουσίαση για την ε, έκθεση του προγράμματος του περιβάλλοντος του ΟΗΕ που θα ασχοληθεί με την ε, απομάκρυνση της οικονομίας από τον άνθρακα. Και βεβαίω εκεί πέρα θα είναι και η κυρία Κονιχέντεγκαρτ για να μας πει τα φιλοδοξία ε, φιλοδοξιών μας. Επίσης θα συνεχίσουμε αυτή την συζήτηση στο υψηλότερο επίπεδο σε άτυπο πλαίσιο στη Βουδαπέστη στο Υπουργικό Συμβούλιο και είπε η Επίτροπος χρειάζεται μια αλλαγή παραδείγματος και εμείς το ίδιο θεωρούμε και ελπίζουμε πως επί προεδρίας μας θα γίνει αυτό και πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια θετικά σημεία ήδη στο Συμβούλιο του Ιουνίου στον Οδικό Χάρτη και έτσι να προχωρήσουμε περαιτέρω στις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε λοιπόν το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στη Βουδαπέστη τέλος Μαρτίου και το Συμβούλιο του Ιωνίου που θα αποφασίσουν για το θέμα αυτό. Είναι ξεκάθαρο το χρονοδιάγραμμα και εύχομαι καλή επιτυχία στην Ουγγρική Προεδρία. Η κυρία Ρωμάνα Γιόρνταν Σισιλ αλλά μου είπε να συνεχίσουμε. Οπότε περνάμε στους ειδικού. Καλωσορίζω λοιπόν τον καθηγητή Wolfgang Lucht, πρόεδρος του ερευνητικού τομέα κλιματικές επιπτώσεις ε, του Ινστιτούτου Ερευνών για τις Κλιματικές Επιπτώσεις στο Potsdam, ο οποίος ε, θα μας πει γιατί ο στόχος μας είναι δύο βαθμοί Κελσίου και όχι 3 παραδείγματος χάρη. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση γνωρίζουμε πως οι ανθρώπινες εκπομπές ε, αερίων αυξάνουν ε, την θερμοκρασία της γης και δεν φαίνεται πως ε, κάποια στιγμή κορυφώνονται οι εκπομπές αυτές. Οπότε οι τωρινές δεσμεύσεις που υπάρχουν δεν είναι δεσμευτικές και μιλάμε σε μια αύξηση κατά 3,2 βαθμών. Οπότε το να περιοριστούμε στους δύο βαθμούς είναι ένας πολιτικός στόχος και όχι ξεκάθαρα επιστημονικός. Καθώς ε, το όριο για τις τοξίνες ε, δεν είναι κάτι το ξεκάθαρο πέρα από το οποίο υπάρχουν οι κίνδυνοι. Υπάρχει ε, ραγδαία αύξηση των κινδύνων με την αύξηση της θερμοκρασίας. Οι επιστήμονες μπορούν να περιγράψουν αυτούς τους κινδύνους και να περιγράψουν βεβαίως τους κινδύνους στα οικολογικά και αγροτικά συστήματα. Λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, δηλώσεις για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής δείχνουν κάποια αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα αυτή υπονοεί επίσης πως ε, και τα πιο υποθετικά αρνητικά αποτελέσματα δεν μπορούν να αποκλειστούν. Ο στόχος των δύο βαθμών ιστορικά βασίζεται σε τρεις ε, λόγους. Πρώτα απ' όλα ότι ο, η θερμοκρασία της γης δεν θα πρέπει να ξεφύγει από αυτό το οποίο είχε τα τελευταί, τις τελευταίες εκατάδες χρόνια πέρα από την υψηλότερη φυσική διακύμανση που είχε στην μηχανική εποχή. Οπότε λέμε να μείνουμε σε αυτά τα όρια. Δεύτερο επιχείρημα είναι πως εάν ξεπεράσουμε τους δύο βαθμούς θα αυξηθούν οι κίνδυνοι στο περιβάλλον και θα μεταμορφωθεί ο κόσμος. Ίσως να υπάρξει και μια κατάρρευση του συστήματος λειτουργίας της γης ε, μεταξύ 2 και 3 βαθμών και βέβαια αυξάνεται κατά πολύ πάνω από τους 3 βαθμούς και ένα τρίτο επιχείρημα είναι πως εάν αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω από 2 βαθμούς το κόστος ε, προσαρμογής θα αρχίσει να ξεπερνάει το κόστος ε, πρόληψης. Εάν αυξηθούν οι θερμοκρασίες ε, κατά δύο βαθμούς, ε, μιλάμε για πάνω από την ξηρά, γιατί η ξηρά θερμαίνεται περισσότερο από τους ωκεανούς και δεν έχουμε ίσο κατανομή, οπότε θα έχουμε μια αύξηση κατά πάνω από τρεις φορές. Οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν ένταση του υδρολογικού κύκλου, η βροχόπτωση θα αυξηθεί σε όγκο και ένταση, οι αλλαγές θερμοκρασία επηρεάζουν την κυκλοφορία στην ατμόσφαιρα και στους ωκεανούς και πάλι θα ενισχυθεί ο κύκλος της βροχής και αυτή η κίνδυνη εμφανίζεται με θερμάτιση πάνω από 2 βαθμούς. Η αύξηση στη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα οδηγήσει σε οξύνηση των ωκεανών, κάτι το οποίο βεβαίως θα δημιουργήσει προβλήματα σε πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς και βεβαίως μπορεί να υπάρξει σε διάφορες καταστάσεις το σύστημα της γης και μπορεί να μεταβεί μεταξύ αυτών των καταστάσεων καθώς θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια σημεία μεταβολής. Ε, η κλιματική ιστορία δείχνει πως υπάρχουν, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι ακριβώς τα όρια. Έχουμε έτσι άρα τυχές κυκλοφορίας των ωκεανών, σταθερότητα των μουσώνων ε, και των ε, στρωμάτων των πάγων. Και βέβαια ο αυξάνεται αν η θέρμανση πάει πάνω από τους δύο βαθμούς. Επίσης, οι ε, πάγοι της ε, Αρκτικής αναμένεται να εξαφανιστούν τελείως τα καλοκαίρια εάν προχωρήσουμε πάνω από 2,5 βαθμούς Κελσίου. Εάν μείνουμε στους δύο βαθμούς, ε, έχουμε μία αύξηση το 2100 του στάθμης θάλασσας κατά 0,8 μέτρα. Επίσης, το υπάγει της Γρυλανδίας, οι οποίοι θεωρούσαμε ότι δεν θα λιώσουν ε, εάν ε, δεν φτάσουμε πάνω από τους 2 βαθμούς, θα μπορούσαν να αρχίσουν να λιώνουν σε μια θέρμανση 1,3 με 3 βαθμούς. Αν φτάσουμε λοιπόν σε 2 βαθμούς θα τελειπωθούν πάρα πολλά οι οικοσυστήματα λόγω, λόγω των αλλαγών στις βροχοπτώσεις και έτσι θα έχουμε προβλήματα με τη βιοπικιλότητα και άρα πάρα πολλά θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν εξαφάνιση. Νέε έρευνε δείχνουν πως υπάρχει ένα σοβαρό κίνδυνος ξύρανσης ε, της λεκάνης του Αμαζονίου σε συνδυασμό με την ε, ανθρώπινη δραστηριότητα. Και αυτός ο κίνδυνος είναι σοβαρότερο στου τρει βαθμού. Ε, Πρόσφατε έρευνε δείχνουν πως τα δάση του Καναδά και της Σιβηρίας κινδύνουν να χάσουν ε, πάρα πολλά δέντρα τους λόγω καλοκαιρινών ξηρασιών και πυρκαγιών που θα προκύψουν και βεβαίως δεν μιλάμε για περίπτωση μαζονίου αλλά αρκετά σοβαρέ στις κοινωνίες μιλάμε κυρίως για το πώς θα αντιμετωπίζουν τις ζέστες του καλοκαιριού την αλλαγή των βροχοπτώσεων και τη μείωση της αγροτικής παραγωγικότητας, ειδικά στους τροπικούς. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια πράγματα ακόμα. Πρώτα απ' όλα, η επιστημονική αβεβαιότητα που υπάρχει ακόμα στις δηλώσεις και κάποια ασάφεια σημαίνει πως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και τα χειρότερα σενάρια. Γιατί η αβεβαιότητα σημαίνει πως δεν μπορούμε ακριβώς να αποκλείσουμε και αυτά τα σενάρια. Επίση, το κόστο προσαρμογή μπορεί να είναι εξίσου μεγάλο με αυτό τη αντιμετώπιση, γιατί απαιτεί διαρθρωτικέ αλλαγέ. Τρίτον, κάποιοι λένε πω ο στόχο των δύο βαθμών είναι ακόμα πολύ επίοικη και πρέπει να πάμε στον 1,5 βαθμό. Κάτι το οποίο βεβαίω θα ευνοήσει τι χαμηλέ περιοχέ, τι νήσου, τι περιοχέ τη Αρκτική και τι φτωχότερε χώρε. Τέταρτον, οι τωρινές προβολές μιλούν για μία ε, ψή, ψήξη λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Αν φύγει αυτή η ατμοσφαιρική ρήπανση θα έχουμε περαιτέρω θέρμανση. Τέλος, οι σημερινές αποφάσεις ε, θα επηρεάσουν το κλίμα σε, στο απότερο μέλλον και έκτον βεβαίως ε, η ακριβής έκταση είναι κάτι το μη ακριβέ. Δηλαδή μπορεί τελικά να είναι λιγότερο αλλά και περισσότερο από δύο βαθμούς, οπότε πρέπει να, να εφαρμόσουμε την αρχή της προφύλαξη. Και τέλος, εάν φτάσουμε σε, δι... σε αύξηση πάνω από δύο βαθμούς από την προβιομηχανική εποχή, έχουμε περάσει σε νέες ανεξερεύνητες ε, περιοχές. Και δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο στο παρελθόν και είναι μάλλον απίθανο το ότι και οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν θα περάσουν σε άγνωστες καταστάσεις. vielen Dank, äh, Professor Lucht, für äh, diese Präsentation. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά για την παρουσίαση αυτή. Σημαίνει δηλαδή δύο Βαθμού Κελσίου. Περνάμε στον δόκτωρα Νίκολα Σένε από την ΕΚΟΦΙΣ, το Ινστιτούτο ΕΚΟΦΙΣ, θα μας αναπτύξει τις μακροοικονομικές επιπτώσεις ε, της και της κλιμάκωσης προς τον στόχο 30%. Σας παρακαλώ να περιοριστείτε σε ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω τα θέματα αυτά. Θα καλύψω τρεις ερωτήσεις. Πρώτη, ε, ε, ποιο είναι το, μερίδιο, το, το δίκαιο μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, επίσης, ε, εάν συμφωνήσουμε με, αυτήν, ε, με το όριο των δύο βαθμών, τι, τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει, αν θέλουμε να το επιτύχουμε για το 2020, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει μέχρι το 2050 να έχουμε ε, μειώσει στο μισό τις ε, συνολικές ε, εκπομπές και επίσης πώς μπορεί να γίνει η κατανομή, τρίτη ερώτηση, πώς μπορεί να γίνει η κατανομή αυτής, αυτού του προϋπολογισμού μεταξύ των χωρών. Μερικοί λένε ότι θα πρέπει αυτοί που έχουν ιστορικά μεγαλύτερες καταναλώσεις να μειώσουν περισσότερο και αντίστοιχα αυτοί που καταναλώνουν λιγότερο να μειώσουν λιγότερο. Αυτή είναι η ευρία άποψη σχετικά με το τι είναι δίκαιο όσον αφορά την μείωση. Εμείς είμαστε οι υπογραφής ε, της ε, τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης ε, του IPCC και οι συνάδελφοι Μισελ Βανέλτσεν και εγώ συγκρίναμε διάφορες μελέτες και είδαμε ότι οι αναπτυγμένες χώρες, οι βιομηχανοποιημένες χώρες θα πρέπει να μειώσουν κατά 25 με 40% σε σχέση με το 1990 τις εκπομπές μέχρι το 2020. Υπάρχουν βεβαίως και αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν ευρέω βεβαίως χρησιμοποιηθεί στις ε, διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις. Ε, υπάρχουν μεμονωμένες προτάσεις οι οποίες είναι χαμηλότερες ή ψηλότερες, αλλά ο μέσος όρος είναι αυτός. Χρησιμοποιώντας και εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μειώσει κατά 30% με 35%. Στο παράρτημα 1 αναφέρεται το 30%. Στην έκθεση IPCC ε, αναφέρονται τα απαραίτητα σε μακροχρόνιο ε, στόχο για το 2050, δηλαδή 80 με 95% και η μείωση θα πρέπει να γίνει 80% τουλάχιστον ε, σε εγχώριο ε, επίπεδο. Ε, και να σας πούμε ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει να μειωθούν στο 50% οι εκπομπές σε σχέση με σήμερα. Πράγμα αρκετά δύσκολο. Είναι, είναι δεσμευτικός αυτός ο στόχος και θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει μια μείωση στο 80% των εγχώριων στόχων. Ε, κατά την άποψή μας ένα ε, δίκαιο μερίδιο θα ήταν το 30%. Ε, το δεύτερο σημείο, ποια είναι, είναι η σωστή αναλογία ανάμειξης στόχων και πολιτικών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αποτελεσματικότητα και μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου. Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά όσον αφορά την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να βελτιωθούμε. Αν θεωρήσουμε ότι αυτοί οι δύο στόχοι έχουν επιτευχθεί, τότε ε, οπωσδήποτε θα έχουμε μια σχεδόν αυτόματη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου, μας το είπε και η κυρία Επίτροπος προηγουμένως, ε, κατά 25% μέχρι το 2020. Εμείς θα θέλαμε να φτάσουμε στο 30% ε, που κατά την άποψή μας είναι ένας καλός υπολογισμός. Επίσης, εάν εφαρμοστούν ε, και οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές και για την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα τότε ε, οπωσδήποτε θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και όσον αφορά το σύστημα εμπορίας ε, δικαιωμάτων ε, εκπομπών. και επομένως θα έχουμε και καλύτερη, καλύτερη αντιστοιχεία με τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να να μας απασχολήσει ε, είναι το εξής, ε, οι οικονομικές επιπτώσεις ε, του να φτάσουμε πέρα από το 20% για αέρια θερμοκηπίου, ποιες θα είναι. Το κόστος της μείωσης των εκπομπών εξαρτάται από την, από την μέθοδο η οποία έχει χρησιμοποιηθεί. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το μακροοικονομικό κόστος θα είναι 81 δις ε, για το 2020 και αυτό αναφέρουν στην, ε, αναφέρει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της ενώ εάν τα πράγματα συνεχίσουν όσο έχουν θα έχουμε ένα 33 δισεκατομμύρια ευρώ για το, το στόχο του 20%. Εάν θεωρήσει κανείς βεβαίως ότι μπορεί να επιτευχθούν σημαντικά οικονομικά ωφέλη από τα μέτρα ε, ενεργειακής αποτελεσματικότητας, ε, τότε θα μπορούσε να υπάρχει αντιστάθμιση ε, του στόχου του 30% και επομένως δεν θα έχουμε οποιοδήποτε επιπλέον, στόχο, επιπλέον κόστος. Την τελευταία, την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε και από το Ινστιτούτο Ερευνών Κλιματικών Επιπτώσεων του Πότσταμ μια μελέτη η οποία θεωρεί ότι το, τα οικονομικά ωφέλη του στόχου του 30% θα είναι ε, σημαντικά εάν υπάρξει καινοτομία και εφαρμογή της στις νέες αγορές. Ε, όμως υπάρχει και μια άλλη ε, άποψη όσον αφορά τις, μακρο, τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις Δηλαδή, εάν ε, ε, ε, μειώσουμε τις εκπομπές με ταχύ μετά το 2020, έτσι ώστε να επιτύχουμε την μείωση του 80-95% μέχρι το 2050, τότε θα είχαμε και μια, και μια αφαίρεση του αποθέματος... Would be του κατακεφαλήν ε, αποθέματος ε, μέχρι το 2050. Όσον αφορά τώρα την ενεργειακή ασφάλεια, ε, είναι γεγονός ότι μέσω των κλιματικών ε, πολιτικών ε, θα είχαμε λιγότερη χρήση ενέργειας, θα είχαμε λιγότερη χρήση στερεών καυσίμων και επομένως σαφή κέρδη, θα είχαμε επομένως και μείωση των χρημάτων που δαπανώνται για την ενέργεια αλλά και δημιουργία θέσεων εργασίας. Ε, ε, σύμφωνα με την Επιτροπή ε, θα είχαμε περίπου 6 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας. Επίσης η υγεία είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που μπορεί να οδηγήσει και σε σημαντικά οικονομικά εφέλη. Επομένως, ε, οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα αυτά στοιχεία, οι περισσότεροι από αυτούς τους οικονομικούς ε, δείκτες ε, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις από την πλευρά της, των πολιτικών και σωστός υπολογισμός του τι σημαίνει δίκαιο μερίδιο όσον αφορά την κατανομή του κόστους. Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε και θα δώσω τον λόγο στον κύριο Γκάι Τέρνερ, διευθυντή στον τομέα έρευνας για τις αγορές άνθρακα στην Bloomberg ε, New Energy Finance. Και από αυτόν βεβαίως θα θέλαμε να ακούσουμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στο σύστημα εμπορίας ε, αερίων και την αποτελεσματικότητά του. Λοιπόν, έχετε 10 λεπτά. To speak, I hope you can hear me now. Ο τίτλος της παρουσίασής μου είναι αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στο πλαίσιο των στόχων του 20 και 30%. Θα σας μεταφέρω κάποια μηνύματα καταρχήν, μήπως και ξεπεράσω το χρόνο μου και μετά θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Πρώτο ζήτημα. Είναι αποτελεσματικό με το 20-30% το σύστημα. Ναι, είναι η απάντηση, βεβαίως. Το σύστημα αυτό, ETS, είναι αποτελεσματικό, ήταν και το 2008 και το 2009, με 5,5% μείωση κάθε φορά. Και όταν μάλιστα αυξήθηκε η τιμή του άνθρωπου και του πετρελαίου πήγε στα 30 παραπάνω. Η μείωση είχε να κάνει πρώτα απ' όλα με την μείωση της τιμής στον άνθρακα και στον ε, ηλεκτρισμό. Στη συνέχεια, 2008-2009, Α, πριν μιλούσα για το 2007-2008, διορθώνει ο 2008 2008-2009 είχαμε μείωση 11% στο σύστημα. Βέβαια, μείωση αυτή δεν οφείλεται μόνο στο σύστημα αυτό καθ' αυτό, οφείλεται και στην ε, κρίση, την οικονομική ύφεση. Πάντως έχουμε κάνει πολλή έρευνα, ήρθαμε σε επαφή με διάφορες ε, εταιρείες παραγωγής ενέργειας και είπαν ότι τώρα αλλάζουν τις αποφάσεις τους για επένδυση εξαιτίας όχι μόνο των ε, τιμών του άνθρακα των συγκεκριμένων τώρα αλλά και των μελλοντικών. Το θέμα είναι ε, η σχέση κόστους και κέρδους του συστήματος αυτού εμπορίας εκπομπών είναι υποφελής πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το θέμα της διαρροής άνθρακα. Θα έρθω σε αυτό. Πάντως ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα πολιτικής είναι σε τι βαθμό η αγορά άνθρακα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε να οδηγηθούμε σε καινοτομία όσον αφορά τον άνθρακα. Ή η αγορά του άνθρακα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε να υπάρξει μια ε, πιο χαμηλή τιμή και η διαφορά να χρησιμοποιηθεί για επένδυση ώστε να υπάρξει περισσότερη γνώση, έρευνα κτλ. για να χρησιμοποιηθούν για νέε ε, τεχνολογίες. Είναι μια, ένα θέμα που πρέπει κανεί να αποφασίσει. Έπειτα, προσοχή, δεν πρέπει να μιλάμε για το 2020. Πρέπει να μιλάμε για το 2030. Όταν παρουσιάζω την ανάλυση μου θα δείτε ότι για το 2020, ό,τι και στόχο βάλουμε για το 2020, οι επιπτώσεις είναι πολύ μικρές. Το σημαντικό είναι τι θα γίνει μέχρι το 2030. Αυτό είναι το βασικό, ιδιαίτερα για την αγορά άνθρακα. Τέταρτον, η αγορά είναι ένα περίπλοκο στοιχείο. Δεν έχει νόημα να προσπαθείς να τη σχεδιάσεις με κάθε λεπτομέρειες γιατί υπάρχει δράση και αντίδραση επηρεάζεται από την κατάσταση που επικρατεί σε άλλους τομείς, σε άλλες αγορές. Αυτά λοιπόν είναι τα μηνύματα που θα ήθελα να σας περάσω. Τώρα πιο συγκεκριμένα, τι έχουμε κάνει. Έχουμε ένα μοντέλο, ακολουθήσαμε τρία διαφορετικά σενάρια. Το πρώτο έχει να κάνει με το στόχο 20% ε, και το 21% μείωση μέχρι το 2020. 30% ε, ερμηνεύεται με 45% μείωση, γιατί μέσω του ETS, του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών, θα έχουμε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Τρία σενάρια λοιπόν είχαμε. Το ένα, η συνέχιση της γραμμής της μείωσης μετά το 2020 με 21%. Το άλλο ήταν ε, με το 30% για το 2020 και μετά ήταν ε, με τον ίδιο ρυθμό, με το ίδιο επίπεδο με μείωση 34% στην ίδια γραμμή. Έπρεπε επίσης να κάνουμε και διάφορες υποθέσεις για εισαγωγές, για την τιμή της ενέργειας κλπ. Και βέβαια το θέμα της τιμής του άνθρακα μια συγκεκριμένη στιγμή. Γιατί δεν μπορείτε να βάλετε την τιμή ένα συγκεκριμένο χρόνο οι τιμές προβλέπονται με 5 και 10 χρόνια πριν. Αν πάρουμε το στόχο του 21% που συνεχίζεται γραμμικά, το 2020 θα είναι 48 ευρώ ο τόνος η τιμή του άνθρακα. Με 34% στόχο γραμμικό πάμε στα 58 ευρώ τον τόνο. Και με το τρίτο σενάριο έχουμε 90 με 100 το 2020. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ επιθετικός αυτός ο στόχος. Όσον αφορά την μείωση των εκπομπών, πετυχαίνουμε τους στόχους που θέλουμε, αλλά εξαιτία των περιορισμών εισαγωγών οι σημερινές ε, εκπομπές θα είναι λιγότερες. Το σημαντικό, η σημαντική επίπτωση είναι στο τομέα παραγωγής ενέργειας. Από εκεί θα έρθουν οι περισσότερες μειώσεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι το φυσικό αέριο που σας βοηθά να πάτε στο 21% και παραπέρα, σταματάει να φτάνει για να πετύχετε το στόχο του 36% 34% μείωση για παράδειγμα και πιο πέρα. Και αυτό που βλέπουμε την προσωμείωση είναι ότι ενώ βλέπουμε αύξηση του φυσικού αερίου που μπορεί να βοηθήσει στην ασφάλεια εφοδιασμού αρχίζει να αντικαθίστεται από λιγνίτη και άλλα. Οι ανανεώσιμες ε, επίσης και εκεί βλέπουμε αλλαγή. Αλλά είναι σημαντικό να δει κανείς πόσο λίγο συνεισφέρει τελικά το φυσικό αέριο στην επίτευξη του πιο μεγάλου στόχου. Και θα σταματήσω γιατί νομίζω ότι εδώ πέρασα το χρόνο μου. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, λέει πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο καθηγητής Μάικλ Κρουπ. Θα μας μιλήσει για την διαρροή άνθρακα. Παρακαλώ. push the button. Pardon. First to the movement of industrial. Αυτό το οποίο λέμε διαρροή άνθρακα είναι η μετατόπιση μηχανικής παραγωγής στο εξωτερικό και εγώ θα ξεκινήσω με ένα παράδοξο για την κλίμακα του προβλήματος. Αν το δούμε με μακροοικονομικούς όρους είναι αμεληταίο. Μιλάμε για λιγότερα από 1% του ΑΕΠ θα μπορούσε να μετακινηθεί. Όσον αφορά το περιβάλλον, είναι κάτι το μέτριο. Μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό των ευρωπαϊκών εκπομπών, αλλά για μερικούς βασικούς τομείς νομίζω είναι κάτι το δυνητικά σημαντικό και όσον αφορά βεβαίως το σχεδιασμό και την πολιτική ανάπτυξη αποτελεσματικού ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας είναι κάτι το κρίσιμο. Και η ανησυχία μου είναι πως η δομή της τωρινής απάντησης θέτει την ευρωπαϊκή βιομηχανία αντίθετη με οποιαδήποτε ενίσχυση κλιματικών στόχων με τρόπους που δεν είναι απαραίτητη. Δεύτερον, το ζήτημα θα έπρεπε να είναι ε, να το δούμε υπό την, ε, το πρίσμα ορισμένων συγκεκριμένων κλάδων και για έναν μόνο από αυτούς πρέπει να δούμε τα πράγματα εκ νέου στη φάση 3. Πριν είχαμε βρει 6-7 τομείς ε, όπου υπήρχε μια πιθανή ανησυχία. Νομίζω για τα σενάρια τιμών κάτω του 30% δεν θα μιλάμε για μεγάλη ε, διεύρυνση. Μιλάμε για τις βασικές, ενέργειες, ε, για τις βασικές βιομηχανίες έντασης ενέργειας. Εγώ μπορώ να μιλήσω επαρκώς μόνο για τρεις κλάδους που έχουμε μελετήσει εις βάθος. Το αλουμίνιο είναι το πιο πολύπλοκο, καθώς θεωρείται αντιπροσωπευτικό όλων των τομέων έντασης ηλεκτρισμού και αυτή τη στιγμή δεν νομίζω πως έχουμε κάποια καλύτερη λύση α, πέραν των όσων προτείνονται. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες. Είναι περίπλοκο αλλά έτσι πρέπει να είναι. Οπότε θα περιοριστώ στο τσιμέντο και το χάλιβα. Κάποιοι θεωρούν πως είναι βαρετά πράγματα, αλλά να σας πενθυμίσω πως αυτοί οι δύο κλάδοι είναι μαζί πάνω από το 1 τρίτο όλων των ευρωπαϊκών βιομηχανικών εκπομπών. Ο καθένας από αυτούς είναι παραπάνω από την αεροπορία ε, και οι δύο μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι, έχουν πενταπλάσει εκπομπές από την αεροπορία και αν σκεφτείτε το πώς ασχολούμαστε με την αεροπορία νομίζω πως πιο στοχευμένη προσέγγιση αξίζει να γίνει σε αυτούς τους τομείς. Θα ξεκινήσω με το τσιμέντο, γιατί είναι το απλούστερο, σαφέστερο και σημαντικότερο. Γιατί? Εν μέρη γιατί είναι σαν τον ηλεκτρισμό, αλλά όχι ακριβώς. Το διεθνές εμπόριο στο τσιμέντο είναι μικρό γιατί είναι βαρύ, κοστίζει μεταφορά του, ειδικά διαξηράς, αλλά είναι επίσης μακράν το αγαθό εκείνο το οποίο είναι έντασης άνθρακα και θα πρέπει να υπάρξει μια υψηλή τιμή για να ξεπεράσουμε το κόστος μεταφοράς. Αναγνωρίζοντας αυτό το πρόβλημα, λοιπόν, η πρόταση είναι να δοθούν δωρεάν άδειες σε όλα τα εργοστάσια παραγωγής, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται και άρα το εάν αντιμετωπίζουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα και να εισαχθούν βεβαίως κάποια αποθέματα για να μπουν νέοι στον κλάδο. Δυστυχώς το τσιμέντο βεβαίως είναι ο κλάδος εκείνος που έχει τη λιγότερη ένταση κεφαλαίου με αποτέλεσμα με τις τιμές που κοιτάμε να είναι επικερδές ε, να είναι κανείς σε μια απόσταση 100 χιλιόμετρα από ένα λιμάνι, να πουλήσει τις άδειες και να εισάγει μετά το τελικό προϊόν. Οπότε θα έχουμε πάλι διαρροή ε, άνθρακα. Οπότε οι αποφάσεις του Δεκεμβρίου για να το αντιμετωπίσουν αυτό έχουν πάλι μια νέα ρήτρα για προσαρμογές εξ Ο αριθμός των αδειών θα μειωθεί αν λειτουργήσει τα κάτω του 50% το εργοστάσιο. Εμείς λέμε πως δεν έχουμε τέτοιες άδειες εξπόστ. Αντιλαμβάνουμε γιατί υπάρχει αυτή η ρήτρα. Βεβαίως, με όλα αυτά τα πράγματα έχουμε εξουδετερώσει τα περισσότερα κίνητρα για να γίνουν πιο αποτελεσματικά τα εργοστάσια τσιμέντου. Τέλος, επειδή παραμένουν προστατευμένα τα εργοστάσια εκείνα τα οποία είναι στην ενδοχώρα, θα δουν πολλά κέρδη. Οπότε θα έχουμε και διαρροή και έκτακτα κέρδη. Για να ξεκινήσω λοιπόν τη συζήτηση με τους συναλληλούς από τη βιομηχανία, εγώ θα έλεγα πως το επίπεδο είναι γύρω στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ στη φάση 3. Οπότε, Ε, προφανώς αυτό είναι προβληματικό από πλευρά σχεδιασμού και συνοψίζω θα μπορούσαμε να έχουμε έκτακτα κέντρα για τις βιομηχανίες, διαρροή άνθρακα και ένα περίπλοκο σύστημα χωρίς κίνητρα και πάρα πολλούς επιθεωρητές. Ε, δεν το θα αυτό. Δεν θέλω να ακουστώ αφελής, αλλά υπάρχει μια πλούστερη ε, λύση, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε το τσιμέντο όπως το πετρέλαιο. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης ε, και να χρειαστεί να αγοράσουν άδειε κτλ. Είναι απολύτω συμβατό με τον ΠΟΕ. Έχουμε πολλές συζητήσεις μαζί τους. Μας είπαν πως δεν θέλουν ε, να μπλέξουν σε τέτοια ιστορία από πλευρά ΠΟΕ, να κατηγορηθούν ότι εμποδίζουν κάποια πολιτική και άρα μπορούμε να επιβάλλουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα αφήσω κατά μέρο. το χάλιβα. Είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποια βεβαιότητα για το εάν χρειαζόμαστε νομίζω κάτι ιδιαίτερο. Αλλά υπάρχει ένα βασικό στρατηγικό ζήτημα με το οποίο θα ήθελα να καταλήξω. Αν θέλουμε κάποιες περιοχές να μπορούν να προχωρήσουν με πιο φιλόδοξους στόχους, και αναμένουμε βεβαίως να χρεώνουν την παραγωγή αλλά όχι τις εισαγωγέ, αυτό γίνεται. Αν περιμένουμε να εξαιρέσουν οποιονδήποτε απειλήσει να μετακινηθεί, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα σοβαρά. Δεν βλέπω προοπτική πολιτική ρεαλιστική να πάμε σε ισχυρότερες λύσεις. Οπότε θα πρέπει τουλάχιστον να ξεφύγουμε από το χάλι που έχουμε στο τσιμέντο. Και βεβαίως αναγνωρίζω πως ο βασικός ε, φόβος βιομηχανίας είναι πως το 30% θα επιδεινώσει την κατάσταση, εγώ θα έλεγα πως είναι μια ευκαιρία να πάμε σε μια καλύτερη πολιτική για να χαράξει τον δρόμο ο κλάδος αυτός και για τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ κύριε Μάικλ Κραμπ. Οπότε, ακούσαμε τις εξαιρετικές παρουσιάσεις και τώρα έχουμε μισή ώρα για ερωτήσεις. Θα δώσω λοιπόν πρώτα απ' όλα τον λόγο στη Γιορτάνα Ευχαριστώ, Τζο. Καλό απόγευμα, κύριε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη για την αργοπορημένη μου αύξηση, αλλά στην Επιτροπή μου, στην Ήτρα, έχουμε Έχουμε ψηφοφορίες και ξέρετε ότι εδώ στο Κοινοβούλιο λέμε πάντα ότι οι ψηφοφορίες έχουν προτεραιότητα. Δυο λόγια να πω έτσι ώστε να ξέρετε τι συμβαίνει και στην Επιτροπή Ήτρε. Γιατί πρέπει να πούμε ότι στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής η πολιτική αλλαγή ε, κλίματος αντιμετωπίζεται όχι μονάχα ως πρόβλημα αλλά και σαν πρόκληση ε, σε σχέση και με την βιομηχανική πολιτική για την πολιτική μεταφορών και πολλών άλλων ε, κλάδων. Επομένως έχουμε δύο επιτροπές οι οποίες είναι υπεύθυνε για το θέμα. Ε, και αυτό ε, σημαίνει ότι το θέμα του άνθρακα θα ειδωθεί από πολλές ε, πλευρές και με σωστό τρόπο. Έχουμε οργανώσει και δύο ακροάσεις, μία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και η δεύτερη θα οργανωθεί από την Επιτροπή Ήτρε στις 17 Μαρτίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 και σας ε, προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την ακρόαση αυτή. Το προσχέδιο της έκθεσης σεισμού ή της γνωμοδότησής μου μάλλον έχει ήδη προετοιμαστεί και βάση της αποτέλεσε, ε, του, αποτέλεσαν οι ήδη υφιστάμενοι κλιματικοί στόχοι για το 2020 στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Θέλουμε σταθερότητα και αξιοπιστία και γνωρίζουμε όλοι ότι θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές μας και από ό,τι ακούω 20% ε, ε, μέχρι ε, το 2020 20 και ακόμα περισσότερο μετά. Ακούγοντας όλα αυτά, ε, που συζητώνται εδώ, ε, είπα στον εαυτό μου τι θα κάνουμε. Πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το σωστό νούμερο. Είναι 24, είναι 25, είναι 30%. Πρέπει να βρούμε ε, ένα συγκεκριμένο ποσοστό και να βρούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι δεν λειτουργούν και που επομένως θα πρέπει να αντικατασταθούν με νέους μηχανισμούς, με νέα εργαλεία έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας να μην χάνουμε όμως χρόνο ε, με αριθμούς και στοιχεία, να προσπαθήσουμε να βρούμε ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία για να επιτύχουμε τους στόχους. Ε, η Επιτροπή Ήτρε πρέπει να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα, μεταξύ αυτών, ας πούμε, τι σημαίνει ότι το κόστος της ε, μείωσης ε, των εκπομπών είναι χαμηλότερο από ό,τι πριν από την οικονομική κρίση. Εγώ βλέπω ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα ε, από ό,τι πριν από την κρίση. Δεύτερον, η μετατόπιση της έδρας των επιχειρήσεων ήδη γίνεται και αυτό βασίζεται στο ETS, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Επίσης, η ενεργειακή αποτελεσματικότητα Εάν έχουμε ε, ήδη, είμαστε ήδη στο σωστό δρόμο, γιατί δυσκολευόμαστε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Επίσης, πώς μπορούμε να κινητροδοτήσουμε τις εταιρείες έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα γιατί είμαστε τόσο μακριά από το στόχο της ε, σωστής ε, χρηματοδότησης ε, των αλλαγών και πώς μπορούμε να κινηθούμε με ταχύτερο ρυθμό προς αυτήν την οικονομία που θα έχει χαμηλή χρήση άνθρακα. Πολλά είναι τα ερωτήματα, τώρα σας έθεσα ορισμένα μεταξύ αυτών. Το θέμα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχουμε ε, και δεν... Ε, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει απλώς να περιοριστούμε σε επιτυχή έκβαση των εσωτερικών μας πολιτικών. Θα πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να είναι θετικές οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε ε, πολύ. Ξέρουμε ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ ε, Ρωμάνα στις ε, συζητήσεις και στις διαδικασίες για την οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακα και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Πέντε ερω... πέντε γεγραμμένοι από ό,τι βλέπω. Ελπίζω να είναι πάρα πολύ σύντομοι ο καθένας από τους εμπειρογνώμονες, ε, ένα λεπτό ε, στον καθένα και ο καθένας από τους εμπειρογνώμονες θα απαντήσει στην ερώτηση που του απευθύνουν οι ε, αγορητές. Ένα λεπτό είναι πάρα πολύ λίγο, λέει ο κύριο Ταταρέλα, εν πάση περιπτώσει εάν σε αυτές τις συνεδριάσεις και συναντήσεις λέμε όλοι ότι ε, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος εάν είχε λιγότερες εκπομπές ε, αερίων. Βεβαίως ε, θα συμφωνούμε όλοι και δεν θα είναι μακριά από έναν επίγειο παράδοσο. Αλλά αυτό είναι της μυθοπλασίας λίγο θέμα και όχι της πολιτικής. Η πολιτική ασχολείται με εργαλεία. Επομένως, συγκεκριμένη απλή ερώτηση. Αν μαζί με τους στόχους ε, δεν θα ήταν πιο χρήσιμο να καθορίσουμε ε, και τα μέσα, τα εργαλεία, τις μεθοδολογίες, τις στρατηγικές, ε, τις τεχνολογίες και τις έρευνες επί των οποίων θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι έτσι ώστε να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ε, οι χώρες ε, οι οποίες ε, μολύνουν περισσότερο είναι αυτές οι οποίες δίνουν και περισσότερα χρήματα στην έρευνα. Δεν θα πρέπει επομένως να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να έχει αποτέλεσμα η έρευνα αυτή τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Ενδιαφέρουσα η άποψή σας. Ναι, αλλά αυτό που λέτε περισσότερη έρευνα, περισσότερα εκπομπές, ναι, ενδιαφέρον. Λοιπόν, Βιτόριο Πρόντι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Το σχέδιο ένα είναι να έχουμε ένα σύστημα ελέγχου των εκπομπών που θα αφορά ολόκληρο τον κόσμο, που θα είναι συνολικό και καθολικό. Για να το επιτύχουμε όμως αυτό πιστεύω ότι και αναφέρομαι εδώ ε, και στα όσα μας είπε ο Δόκτωρ Τέρνερ, θα πρέπει ε, να το συνδυάσουμε με τον στόχο του να φτάσουμε σε ένα απλό σύστημα. Ένα σύστημα που θα είναι απλό. Πιστεύω ότι το σύστημα της ε, Επιτροπής, το οποίο είναι κατακαιρματισμένο και ασχολείται με το μίσ δεν είναι ορθό και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σωστά, γιατί προβλέπει και την δημιουργία ενός ε, ε, ε, συνολικού εργαλείου. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιβάλλουμε τελικά ένα πιο απλό σύστημα το οποίο θα φορολογεί στην πηγή όλα τα στερεά καύσιμα και όχι κατά, τμήματα γιατί διαφορετικά, όπως έχουμε τώρα δηλαδή, γιατί διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει σωστά η αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very uh, Ευχαριστώ πολύ. Είπατε, κύριε καθηγητά, ότι έχετε μια ιδέα για έναν ειδικό τομέα, για το χάλιβα, αλλά ότι δεν είχατε χρόνο να μας πείτε περισσότερα. Μήπως μπορείτε παρόλα αυτά, απαντώντας στην ερώτησή μου, να μας εξηγήσετε τι εννοούσατε, ποια ήταν αυτή η ιδέα σας. Ευχαριστώ, Ρίτσαρτ Σέβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να σχολιάσω αποκαλυπτικές απόψεις, όπως αυτές που ακούσαμε εδώ. Έχω όμως την εντύπωση ότι καλούμεθα να ενισχύσουμε τον μηχανισμό εμπορίας δικαιωμάτων. Όμως έτσι δημιουργούμε μια τεχνητή αγορά. Και τελικά αυτοί που την κατακρίνουν αυτή την τεχνητή αγορά είναι αυτοί που την δημιούργησαν. Το βασικό ζήτημα είναι πώς ε, θα φτάσουμε στους δύο βαθμούς. Εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνει εύκολο, ακόμα και αν πάμε από το 20% στο 30% γιατί υπάρχουν χώρες όπως είναι η Κίνα που δεν έχουν όριο, δεν έχουν ε, τους ίδιους περιορισμούς όπως αυτοί που βάζουμε εμείς. Οπότε τι άλλες δυνατότητες βλέπει η επιστήμη προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές χωρίς να περάσουμε από το 20% στο 30%. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. ευχαριστούμε τώρα. Δύο ερωτήσεις έχω. Στον Τέρνο πρώτα απ' όλα. Στον Τέρνο και στον Κράπ. Στους δύο καθηγητές. Εκτός από το ETS υπάρχουν άλλα μέτρα, κάποια dividend για παράδειγμα, όπως λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δίνεται κάποιο μερίδιο στον πληθυσμό. Ναι, οι εταιρείε ε, πληρώνουν το κόστος, αλλά μετά αυτό κατανέμεται στον κόσμο. Μήπως είναι ένας καλός τρόπος αυτός για να βοηθήσουμε να απαλλαγούν από την ενεργειακή εξάρτηση οι άνθρωποι και προς τον κύριο Χένε. Αν θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές, από την άλλη μεριά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι η ανεργία στις χώρες μας. Πέρυσι 0,7% ήταν ε, η ανάπτυξη. Εσείς βλέπετε κάποιο σενάριο το οποίο να συμβιβάζει ε, το πρόβλημα που έχουμε με την ανεργία, δηλαδή να μην χαθούν και άλλες θέσεις απασχόλησης με ε, την μείωση των εκπομπών. Να συμπληρώσω κι εγώ λίγο. Για το 20% το στόχο αυτό, 20%. Είπατε ότι βοηθάει, αλλά όχι το 30%. Δηλαδή λέτε ότι για το φυσικό αέριο ότι δεν είναι αυτό που θα βοηθήσει περισσότερο. Μετά προτείνατε είπατε ότι το 30% ότι θα προχωρήσουμε στο λιγνίτι. Αυτό είπατε, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα καλά. Έπειτα για το τσιμέντο, βιομηχανία. Λέτε ότι η πολιτική μας που δίνει δωρεάν δικαιώματα στην ε, βιομηχανία θα είναι αποτυχία, αυτό λέτε. Και τι προτείνετε ως εναλλακτική λύση για την τσιμεντοβιομηχανία. Uh, Ο κύριος Εχουάουτ προς τον κύριο Λιούχ θέλω να ρωτήσω κάτι. Θα υπάρξει το 2014 μια έκθεση από τα EPCC. Τι περιμένετε εσείς, ποια περιμένετε ότι θα είναι η κατεύθυνση των συμπερασμάτων της έκθεσης αυτής στον κύριο Χένε, τον δόκτωρ Χένε. Μπορείτε να μας μιλήσετε περισσότερο για το δίκαιο αυτό μερίδιο ε, για το οποίο μιλήσατε ανάμεσα στο σύστημα εμπορίας ε, και εκτός συστήματος εμπορίας. Άλλη ερώτηση προς τον κύριο Τέρνορ. Για τις τιμές του άνθρακα, στις οποίες αναφερθήκατε και είπατε ότι επηρεάζουν. Έχετε, δείτε, έχετε δει μήπως τι τιμές χρειάζονται για το μέλλον ώστε να επηρεάσουν κάπως τα πράγματα μετά από το 2007 και 2008, από αυτά που ξέρετε δηλαδή βάσει της εμπειρίας σας. Τέλος το για καθηγητή Κραπ. Είναι ξεκάθαρο ότι το σημερινό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων δημιουργεί προβλήματα. Εντάξει, η Κομισιόν προσπαθεί να βρει κάποιες δυνατότητες να τα διορθώσει χωρίς να γίνουν τεράστιες αλλαγές στο τρέχον σύστημα. Για παράδειγμα, μειώνοντας τα δικαιώματα. Εσείς μπορείτε να σχολιάσετε την προσέγγιση αυτή της Κομισιόν. Έχουμε ακόμα δύο-τρεις ερωτήσεις. Αλλά να ρωτήσω εγώ. Είπατε ότι δεν είναι το 2020 αλλά το 2003. Ενώ ο καθηγητής Τέρνερ είπε ότι πριν από το 2020 θα φτάσουμε στο αποκορύφωμα. Τελικά, τι ισχύει, 2020 ή 2030 ποια δεκαετία είναι η πιο σημαντική. Αυτή η επόμενη, γιατί αυτό πρέπει να το ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι. Έχουμε χάσει χρόνο ή μπορούμε να περιμένουμε ακόμα μέχρι το 2030. Για τη Χαλιβουργία επίσης θέλω να ακούσω περισσότερα. Ο κύριος Χροπ θα ήθελα να μας πει μερικά περισσότερα πράγματα για τη Χαλιβουργία, πού βρισκόμαστε ακριβώς. Και επί τόπος και Μακάβεν, έτσι και εγώ δεν έχω καταλάβει, Αυτά φτάσουμε 34% μείωση, τι εννοούσατε με το λιγνίτι, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα. Εμείς θέλουμε ανανεώσιμες, δεν θέλουμε άνθρακα λιγνίτι. Δεν σας κατάλαβα εκεί. Μας είπατε ότι είμαστε στο, σωστό δρόμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε περισσότερο, οπότε θα έχουμε προχωρήσει περισσότερο από το 20% για το 2020. Έτσι δεν είναι και άρα θα έχουμε περιθώριο λιγμών. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μας λοιπόν. Με αυτές. Παρακαλώ. Ναι, και εγώ για το χάλιβα ήθελα να ρωτήσω. Ωραία, βλέπετε ότι πολύ ενδιαφερόμαστε για το χάλιβα εδώ. Οπότε ας ξεκινήσουμε με τις απαντήσεις. Σύντομα παρακαλώ. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. αναφερθήκατε στην πέμπτη εκτίση αξιολόγησης του IPCC Κοιτάξτε, ολοκληρώθηκε τώρα, αλλά θα υπάρξουν και κάποιες ειδικέ ε, ε, εκθέσεις έτσι ώστε να, που θα κυκλοφορήσουν μέχρι το καλοκαίρι έτσι ώστε να καλυφθούν κάποια κενά. Ε, στην επόμενη αξιολόγηση για το 2014 ε, θα εστιάσουμε σε τρία πράγματα. Πρώτον, ε, θα έχουμε καλύτερη ακόμα βάση όσον αφορά τις, τα, τα επιστημονικά συμπεράσματα, γιατί η βάση εργασίας είναι καλύτερη. Δεύτερον, το, όλα τα ζητήματα θα ειδωθούν σαν ένα κομμάτι ε, ενός γενικότερου πλαισίου ε, σταθερότητας που δημιουργείται πλέον. Τρίτον, τρίτον είναι ακόμα πρόημο, αλλά ελπίζω ότι ε, το κόστος, ότι θα υπάρχει καλύτερη, προσαρμο, ε, καλύτερη ε, διασύνδεση ανάμεσα στο κόστος προσαρμογής και το κόστος πρόληψης. Και νομίζω ότι όσον αφορά τα, τις οδούς που θα πρέπει να ακολουθηθούν για το αποτέλεσμα που θέλουμε, θα έχουμε καλύτερες εναλλακτικές λύσεις. Ε, τώρα είπατε ότι είναι ουτοπία αυτό που λέμε, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ε, ότι μπορούν οι στόχοι να επιτευχθούν μέχρι το 2050 ε, και ορισμένα αποτελέσματα έχουν ήδη επιτευχθεί και όσον αφορά τον προϋπολογισμό την πρώτη δεκαετία και επομένως τα επόμενα 20 χρόνια και τα άλλα 20 μέχρι το 50 μπορούμε, το 2050 μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα έχουμε επιτυχία. Εν πάση περιπτώσει, αν ληφθούν τώρα κάποια μέτρα θα είναι πολύ καλύτερο. Όσον αφορά τα σενάρια τα οποία βασίζονται πάντοτε στην ε, ανάπτυξη, ε, πιστεύω ότι έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά τον έλεγχο ε, του υλικού, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με την εξόριξη, με την, με την εξόριξη πρώτων υλών, με την βιομάζα, με τον υπολογισμό της αλλαγής επιφάνειας. Ναι, βεβαίως υπάρχουν και νέα στοιχεία όσον αφορά τον ε, υπολογισμό και πάντα το ερώτημα είναι ε, πόσος είναι ο όγκος των στοιχείων. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό, την αύξηση του, του πληθυσμού. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία, τα παράμετροι που αλλάζουν και βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν όλες αυτές οι παράμετροι υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δόκτωρ Ευχαριστώ πολύ. Ε, στο ερώτημα αν μπορούμε να περιμένουμε τώρα και να ε, προχωρήσουμε λίγο αργότερα. Υπάρχουν ε, σενάρια τα οποία δείχνουν την τωρινή δέσμευση των χωρών στη διαδρομή από την Κοπεϊχάγη στην Κανκούν και ακόμα πιο πέρα. Νομίζω ότι εάν έχουμε μετριοπαθείς, κάνουμε μετριοπαθείς προσπάθειες τώρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και εν πάση περιπτώσει σίγουρα πολύ δαπανηρό ε, να επιτύχουμε τους στόχους μας ε, αργότερα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως ε, τονίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τώρα. Σχετικά με την δυνατότητα της αύξησης, της επίτευξης του στόχου του 2% χωρίς αύξηση από το 20 μέχρι το 30, ναι θα μπορούσε να είναι δυνατόν, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αντισταθμίσεις σε, εθνικό, σε διεθνές, συγγνώμη, σε παγκόσμιο ε, επίπεδο εάν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήσει τις φιλοδεξίες της ενδεχομένως και κάποιες άλλες χώρες να μπορούν να το κάνουν αλλά υπάρχουν και χώρες όπως η Κίνα η Κίνα ε, προχωράει και θα με μεγάλη ε, προσμονή θα περιμένω να δω το πενταετές πρόγραμμα της Κίνας ένα άλλο ζήτημα όσον αφορά ε, την, ε, το σωστό, το ορθό δίκαιο μερίδιο ανάμεσα στο κόστος προσαρμογής και το κόστος ε, πρόληψης, εμείς πιστεύουμε ότι εάν εφαρμόσει κανείς και τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους στόχους για την ενεργειακή αποδοτικότητα, τότε μπορεί άνετα να φτάσει στο 40% χωρίς πρόβλημα. Όσον αφορά το συσχετισμό ανάμεσα στις πολιτικές ε, και τους ε, αριθμούς ε, πιστεύω ότι και τα ποσοστά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για την βιομηχανία να μην ακολουθήσει αυτά τα προγράμματα. Είναι σαφές αυτό. Ο κύριος Τέρνερ. Για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. εάν ε, ε, θα μπορέσουμε στη δεκαετία 2030 να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Εγώ θα προτιμούσα να μην περιμένουμε, να ξεκινήσουμε συγκεκριμένα βήματα από τώρα. Εάν ε, η στρατηγική είναι ελκυστική, τότε οπωσδήποτε θα αντιδράσουν και οι αγορές και θα ακολουθήσουν και οι τιμές. Εάν ενθαρρύνουμε και δώσουμε κίνητρα στις νέες τεχνολογίες, λαμβάνοντας βεβαίως πάντα υπόψη ότι ε, η αγορά γνωρίζει ότι ε, όσο προχωράμε ε, μπορεί να γίνει πιο φτηνή μια, να γίνει πιο φτηνό ένα μέσον και άρα το προβλέπουν οι αγορές. Πάντως Πιστεύουμε ότι ε, χωρίς αμφιβολία θα αυξηθεί η τιμή του άνθρακα σε περίπτωση που οι δύο προηγούμενες ε, προϋποθέσεις ε, δεν αντιμετωπιστούν. στο νέο ETS μπορούν, ε, μπορεί να υπάρξει ε, μειωσία αν χρησιμοποιηθεί τεχνολογία ε, περίπου 6 δις ευρώ και επομένως τα CGDs μαζί με την τροποποίηση των εφαρμογών μπορεί να, γίνει, να καταστήσει το φυσικό αέριο πιο ακριβό στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Και καταλαβαίνουμε ότι εδώ υπάρχει ένα κριτήριο αναφοράς. Αυτό είναι ένα κριτήριο αναφοράς όσον αφορά την ε, ε, τιμή για το νέο ETS. Επομένως, απαντώ λέγοντας ότι θα πρέπει να απλουστεύσουμε το ε, σύστημα. Ε, ήδη έχουμε πολύ σημαντική απλούστευση, αλλά εάν υπεραπλουστεύσουμε το σύστημα, τότε ενδεχομένως θα οδηγήσει ε, σε αποκλήσεις και σίγουρα σε άδικη κατάτμιση των υποχρεώσεων η πτυτικότητα των αγορών, η αστάθεια δηλαδή των αγορών ε, ενδεχομένως οφείλεται στο ότι δεν έχει αλλάξει το ETS το τελευταία, τα τελευταία ε, δύο χρόνια. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί, δεν μπορεί κανείς να τροποποιήσει τις τιμές γιατί έχουν την σταθερότητα που χρειάζονται και νομίζω ότι αυτό το στόχος του 34% για το 2030 για το φυσικό αέριο τότε ε, μπορεί κανείς να επιτύχει το 2% επιπλέον μέχρι το 50% αλλά δεν μπορεί μόνο με το φυσικό αέριο να, να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σκρόπ. Πολλές ερωτήσεις ακούστηκαν για άλλες δυνατότητες, για άλλες πολιτικές και τη σχέση μεταξύ τους. Εγώ δεν έχω δει κανένα πακέτο πολιτικής που να μην περιλαμβάνει συνδυασμό και τεχνολογία και απόδοση ενέργειας και μείωση χρήσης άνθρακα. Ο συνδυασμός εξαρτάται βέβαια και το μείγμα από τον τομέα. Για μένα Πάντως ο συνδυασμός αυτός είναι ό,τι καλύτερο. Για το χάλιβα, επειδή με ρωτήσατε για το χάλιβα, και οι τιμές και οι επενδύσεις στην καινοτομία είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι κάτι που έχει ήδη γίνει στον τομέα κατά πολύ. Συνεπώς, η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι οποιοδήποτε σύστημα καθορισμού τιμών του άνθρακα, είτε πρόκειται για το ETS, είτε πρόκειται για φορολόγηση οτιδήποτε, ποτέ δεν θα έχουμε την ίδια τιμή σε όλες τις περιοχές συγχρόνως. Είναι ψευδέστηση να νομίζουμε ότι θα το πετύχουμε, άρα τι μπορούμε να κάνουμε ή που θα βγάλουμε την τιμή του άνθρακα από αυτές τι δραστηριότητες, παρόλο που κάναμε πολύ κόπο για να τις εντάξουμε, ή αλλιώ δεν θα υπάρχει διάκριση στους ε, εσωτερικούς παραγωγούς σε σχέση με τους ε, εκτός των χωρών μας. Αυτό που προσπάθησα δηλαδή να πω όσον αφορά το χάλιβα και τη χαλιβουργία είναι ότι η ίδια λογική εφαρμόζεται που λέει ότι τελικά πρέπει να έχουμε ένα σύστημα όπου οι καταναλωτές χάλιβα θα αντιμετωπίσουν ένα σύστημα τιμών, είτε πρόκειται για την εσωτερική παραγωγή, είτε για τις ε, εισαγωγές. Αλλά ότι θα υπάρξει κάποιο αντιστάθμισμα για τη δαπάνη αυτή. Αυτό είναι που λέμε και για το τσιμέντο. Στο χάλιβα είναι θεμητό, είναι κάτι το οποίο συζητιέται από τους ειδικού και τους ερευνητές. Είναι απόλυτα θεμητό να πούμε ότι στο στάδιο 3 πρέπει να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο. Και ο βασικός λόγος που δεν υπάρχει είναι ότι η εντατική βιομηχανία ε, χρειάζονται πολλά χρήματα. Η βιομηχανία χρειάζεται βεβαιότητα και ο μόνος τρόπος είναι όχι να έχουμε πολιτικά παιχνίδια για, για πόσο κρατάνε τα συστήματα εμπορίας και τα λοιπά και τα δικαιώματα, αλλά ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σύστημα όπου δεν θα υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην εχώρια παραγωγή και τις αγωγές. Και η βιομηχανία πιστεύει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε στο τσιμέντο για τους ίδιους λόγους δεν μπορούμε να περιμένουμε Παρόλο που εκεί οι τιμές μπορούν να αυξομοιώνονται χωρίς τόσο μεγάλο πρόβλημα, όταν υπήρχε κατάρρευση στο πρώτο στάδιο, είπαμε γιατί κανείς δεν μας το είπε. Πρέπει να έχουμε ένα συνδυασμό και κέρδους και διαρροής άνθρακα που το κόστος να πηγαίνει σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εγώ στηρίζω απόλυτα το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο σύστημα. Ευχαριστούμε για τον πρώτο αυτό γύρο. Ακούσαμε όλους τους εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο τμήμα μέρος 3 ονομάζεται, αλλά τέλος πάντων από πλευράς εμπειρογνωμόνων είναι το δεύτερο. Θα δώσω το λόγο στον Άξελ Έγκερτ, Διευθυντής Δημοσίων Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιομηχανιών Σιδήρου και Χάλιβα της Eurofair. Και εσείς πρέπει να απαντήσετε στο ίδιο ερώτημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πρόσωπο της Βιομηχανίας Έντασης Ενέργειας. Εγώ προέρχομαι από τη Χαλιβουργία Ελπίζω ο χρόνος να είναι αρκετό. Έχω γύρω 40 σελίδε εντωμεταξύ τη μείωσα. Πρώτα απ' όλα εκπροσωπώ τι βιομηχανίε ένταση ενέργεια. Γυαλί, χαρτί, τσιμέντο, χημικά, δηληστήρια, χάλιβα, μη συντρούχα μεταλλεύματα. Οι βιομηχανίε αυτέ ε, έχουν δεσμευτεί να μειώσουν περαιτέρω τι εκπομπέ του. Πρέπει να το πω αυτό. Δεν είμαστε κατά τη προστασία του κλίματο και α συνεισφέρουμε όσο μπορούμε από τεχνική και ανταγωνιστική πλευρά. Δεν είμαστε κατά του στόχου του 20% αρκεί η διεθνή μας ανταγωνιστικότητα να μην επηρεαστεί περαιτέρω. Πρέπει να αποδεχτούμε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το Συμβούλιο το 2007 και επανέλαβε το 2008 και 2009 για να προχωρήσει στο 30% μόνο υπό τον όρο πως οι άλλες χώρες αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες οικονομίες θα μας ακολουθήσουν. Αυτό προφανώς δεν έγινε ούτε στην Κοπενχάγη ούτε στο Βανκούν. Οπότε, όπως είπε μόλις ο κ. Γκραμπ, πρέπει να έχουμε σταθερότητα. Θέλουμε αυτή την βεβαιότητα. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Να σας δώσω ένα παράδειγμα οι δεσμεύσει ε, της Κίνας ε, να μειώσει κατά 40% κατ' ουσίαν σημαίνει αύξηση εκπομπών από 75% έως 90% μέχρι το 2050. Αυτό τον υπολογισμό κάνουμε. Μιλάμε για ε, αύξηση 52 δισεκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα σε 10 χρόνια. Αυτή η αύξηση μόνο είναι παραπάνω από τις συνολικές εκπομπές της Ένωσης Οπότε θα πρέπει να σβήσουμε όλα τα φώτα στην Ευρώπη και ακόμα δεν θα μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε αυτή την αύξηση. Μόνο την αύξηση. Ίσως καλό θα ήταν η Κομισιόν να κάνει μια τέτοια αξιολόγηση και για άλλες χώρες όπως Βραζιλία, Ινδία κτλ. Τα νούμερο αυτό δείχνει πως δεν μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη αυτή αν δεν γίνουν δεσμεύσεις και από τις άλλες οικονομίες. Δεν έχει νόημα να θυσιάζουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία εάν αυξάνονται οι παγκόσμιες εκπομπές. Οπότε επιμένουμε στις δεσμεύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να περάσω στα μοντέλα που χρησιμοποιεί η Κομισιόν για την αξιολόγησή της. Εμείς θεωρούμε πως τα μοντέλα της Κομισιόν βασίζονται σε κάποιες προκαταλήψεις που υποτιμούν την διαρροή και τις αρνητικές επιπτώσεις στη βιομηχανία και την απασχόληση, υποτιμούν την τιμή του άνθρακα, την αυστηρότητα των ορίων, δεν υπολογίζουν το ότι ήδη οι τιμές του ηλεκτρισμού στην Ευρώπη είναι πάνω από 20% ακριβότερες από τη ΣΥΠΑ και 200% ακριβότερες από την Κίνα, δεν υπολογίζουν το υπεραιτέρω αύξηση της τιμής του ηλεκτρισμού λόγω της εφαρμογής της τρίτης φάσης του ETS, δεν υπολογίζουν την νομοθεσία περί ανανεώσιμων που επίσης ε, θα αυξήσει την τιμή του ηλεκτρισμού. Τα μοντέλα αυτά δείχνουν περιορισμένη επίπτωση στην, ε, στις, ε, στο εργατικό δυναμικό γιατί θεωρείται πως ε, το κόστος από τις δημοπρασίες θα πάει πλήρως στην εργασία, κατά το οποίο δεν σκοπεύουν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Επίση, εμεί έχουμε περιορισμού που δεν έχουν οι ανταγωνιστέ μα, όπω παραδείγματο χάρη κόστο λόγω τη περιβαλλοντική νομοθεσία τη Ένωση, διοικητικό άχθο, άδειε και ακόμη πιο σημαντικό, τα μοντέλα δεν αναφέρουν την, το τι γίνεται με τις επενδυτικές αποφάσεις. Όλα αυτά δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Οπότε τα μοντέλα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και την δυναμική της αγοράς. Η ανακοίνωση υπολογίζει το κόστος ε, του στόχου 30% σε 0,54% του ΑΕΠ. Σε αντίθεση με αυτό, μία έκθεση του Αυστριακού Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας και του Ινστιτούτου Βέγνερ την προηγούμενη εβδομάδα υπολογίζει το κόστος σε 2% του ΑΕΠ. Ήδη για το στόχο 20%. Οπότε τα μοντέλα της Κομισιόν βασίζονται κυρίως στο 20% που προήλθε τη μείωση από την οικονομική κρίση και λένε πως για περαιτέρω μειώσεις θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο 60%. Αλλά αυτό το κάνουμε τα νούμερα του 2008. Γιατί δεν το κάνουμε τα νούμερα του 2010. Τότε θα βλέπαμε πως θα είχαμε μια αύξηση κόστους 69%. Η τιμή του άνθρακα. Τα μοντέλα της Κομισιόν προβλέπει στην τρίτη περίοδο μία τιμή 60 και μισό ευρώ. Εμείς κάναμε αναλύσεις των προβλέψεων για το στόχο του 20% που έχουν δημοσιευτεί από την Barclays, Deutsche Bank, Saga Carbon, Obeo, UBS και άλλες πηγές. Η μέση τιμή του άνθρακα προβλέπεται στα 28 ευρώ και όχι 16,50. Η πρόβλεψη για το 2020 είναι 36 ευρώ. Οπότε σχηματίζεται μια διαφορετική εικόνα από αυτή που μας λέει η Κομισιόν και ήδη αυτή είναι η τιμή που θέλει να επιτύχει η Κομισιόν με το στόχο του 30%. Να μου επιτρέπετε άλλες δύο παρατηρήσεις που θα έπρεπε να σκεφτείτε. Πρώτα απ' όλα, τι θα γίνει αν έχουμε και άλλη κρίση. Θα έχουμε πρόταση να περάσουμε στο 40% μέχρι το 2020. Δεύτερον, θα ανησυχούμε εμείς για καθόλου βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Γιατί αν γίνει αυτό θα χρειάζονται λιγότερες άδειε και θα πέσει η τιμή. Οι εταιρείε βελτιώνουν την απόδοση από το 2008 και πρόκειται για επενδυτικές αποφάσεις προκρίσεις. Παραδείγματο χάρη, έχουμε στην ε, εκλογική περιφέρεια του Προέδρου ένα αέριο βιοαερίου που θα εξοικονομήσει 460.000 τόνους ε, ε, αερίου το χρόνο. Θα τιμωρηθούμε γι' αυτό με υψηλότερους στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Έγκερτ για τις παρατηρήσεις αυτές, ε, για την ανακοίνωση της Κομισιόν. Συνεχίζουμε με την Σαντρίν Ντίξον Ντεκλέβ, Διευθύντρια to the Prince of Wales EU Corporate Leaders Group on Climate Change. Και θα σας ακούσουμε. Παρακαλώ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω εδώ σήμερα. Μιλάω εκ μέρους του Prince of Wales από το Ηνωμένο Βασίλειο και το EU Corporate Leaders Groups on Climate Change, που είναι δύο ε, όμιλοι οι οποίοι ζητούν φιλόδοξους στόχους μείωσης ε, χρήσης άνθρακα και εκπομπών. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε όντως επικοδομητική συζήτηση για τις διαφορετικές στάσεις των επιχειρήσεων. Οι δύο όμιλοι μου πάντως συμφωνούν με την προοπτική υπέρ της ανάπτυξης με μείωση χρήσης άνθρακα πιστεύοντας ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε να μην χάσουμε τις αγορές μας, οι οποίες κινδυνεύουν να πάνε προς την Κίνα της Ηνωμένες Πολιτείες. Συμμετέχουν στους ομίλους αυτούς πολλές εταιρείες από ασφάλειες, τράπεζες, επικοινωνία. Με διάφορα ανακοινοθέντα έχουν υποστηρίξει το διεθνές πλαίσιο με φιλόδοξους στόχους προκειμένου να υπάρξουν κίνητρα για μια οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακα. Τα μέλη μας δεν εκπροσωπούν επιχειρήσεις μόνο καθαρής ενέργειας. Όχι, έχουμε την Deutsche Telekom, την Nissan, τη Philips, την Shell, την Unilever, την Simex, Cimenta, αλλά και την Tesco και άλλες. Όλες αυτές οι εταιρείες τι πιστεύουν. Πιστεύουν ότι πρέπει να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο και ότι αυτό ο ηγετικός ρόλο θα μα φέρει πλεονεκτήματα. Τρία πράγματα πιστεύουμε. Ότι ο μεγαλύτερο κίνδυνος για την Ευρώπη και την ανταγωνιστικότητά τη, είναι να μείνει αδρανή. Ότι η λιγότερη χρήση άνθρακα προσφέρει ωφέλη για το μέλλον και ότι μια κοινωνία που παίρνει χαμηλό κίνδυνο όσον αφορά το κλίμα είναι μια κοινωνία πιο προσιτή προς τους πολίτες της και πιο βιώσιμη. Όπως είπε και η συγκήτρια από την Ήτρε, εμείς θέλουμε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, η οποία να προσφέρει στόχους μείωσης άνθρακα κατά 80 και 95%. Ε, χαιρόμαστε που θα έχουμε τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο έγγραφο. Αυτό ξεκινάει ένα διάλογο για να δούμε ποια είναι η σχέση κόστους και ωφέλους από τη μείωση άνθρακα. Πολύ σημαντικό για να υπάρξει νέα ροή κεφαλαίου και επενδύσεις σε υποδομές χαμηλής χρήσης άνθρακα, μεταφορές, ε, γεωργία κλπ. Όπως ξέρετε, Πρόεδρε, αν και δεν ήσασταν ε, παρόν εκείνη την ημέρα, ήσασταν εκτός της χώρας, είχαμε μια διάσκεψη κορυφής για χαμηλή χρήση άνθρακα με συμμετοχή του Πρόεδρου Παρόσο και του ε, Πρόεδρου Φανερομπάου. Είχαμε και την υψηλότητα των πρίγκιπα της Ουαλίας ε, και πολλούς ε, διάσημους οικονομολόγους και επικεφαλής επιχειρήσεων. Το μήνυμα που βγήκε ήταν ότι μπορούμε να πετύχουμε ε, την ευημερία μας μέσω χαμηλότερης χρήσης άνθρακα, ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, αλλά χρειαζόμαστε φιλόδοξους στόχους και το σωστό πλαίσιο. Ακούσαμε το πεντετές σχέδιο των Κινέζων, αλλά να ξέρετε ότι και άλλες χώρες προσελκύουν επενδύσεις, ενώ εμείς όχι, βρισκόμαστε πολύ πίσω όσον αφορά τις επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες. Είπαμε τότε ότι το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου πρέπει να έρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και υπάρχει, είναι έτοιμο να επενδυθεί. 83 δολάρια στα τέλη του 2008 και μάλιστα σε ένα έτος που είχαμε ύφεση. Παρ' όλα αυτά, επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες επένδυσαν 178 δισεκατομμύρια ευρώ σε ε, καθαρή ενέργεια ανά τον κόσμο. 30% το 2009. Στην ε, Ευρώπη όμως επικρατεί μια έλλειψη εμπιστοσύνη, μια βεβαιότητα για το δρόμο που ακολουθούν οι πολιτικές. Και αυτό το βρίσκουμε στις διάφορες χώρες μας. Και αυτό είναι το οποίο υπονομεύει και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Στη διάσκεψη αυτή αναφερθήκαμε και στους μηχανισμούς και είπαμε ότι οι επίτροποι όσοι αποφασίζουν για τις πολιτικές πρέπει να φροντίσουν να γίνει πραγματικότητα ο στόχος μας. Έχουμε καταλάβει ότι η βιομηχανική ανάπτυξη δεν σημαίνει περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όχι. Μπορούν να συνδυαστούν οι χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με ε, μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη. Όπως και επιχειρήσεις που το έχουν καταλάβει αυτό, έτσι και οι χώρες μπορούν να κάνουν το ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι από την αρχή της δεκαετίας του 90 το ακαθάριστο αθρικό προϊόν μας έχει αυξηθεί κατά 40%. Η παραγωγή μας κατά 30%. Ενώ οι εκπομπές έχουν μειωθεί το 2009 κατά 17,3%. Πολλές εκθέσεις λένε ότι είναι εφικτή η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε ότι μπορούμε να έχουμε επιπλέον 6 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και αυτό είναι κάτι εφικτό πολύ σύντομα, όπως επίσης και η επίτευξη του στόχου μας του 30% για το 2020. Έχετε δίκιο πάντως ότι ο στόχος του 20% είναι πιο κοντά σήμερα εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης. Δεν είναι πρόβλημα πια αυτό. Το αναγνωρίζουμε αλλά δεν φτάνει για να προσελκύσει νέες επενδύσεις στην καθαρή τεχνολογία και στις υποδομές για να πετύχουμε το στόχο του 80 με 95%. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας λέει ότι 20% στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς ε, επιπλέον ε, μειώσεις σε εθνικό επίπεδο από τώρα μέχρι το 2020. Επειδή μπορούμε να έχουμε πολλά ωφέλη από τους στόχους μας για την ενεργειακή απόδοση, γι' αυτό και πιστεύουμε ότι και η μείωση αερίου του θερμοκηπίου θα επιτευχθεί πιο εύκολα. Πάντως, πολύ σοβαρές προσπάθειες από τα κράτη-μέλη για την ενεργειακή απόδοση μπορούν να βοηθήσουν εφόσον συνοδευτούν από απόσυση δικαιωμάτων κατά την τρίτη φάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει, για το οποίο πρέπει να φροντίσουν και οι πολιτικοί σε όλες τις χώρες μας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ μπορώ, μπορώ να σας παρακολουθήσω τουλάχιστον από τα γερμανικά, κάπως γρήγορα. Περνάμε λοιπόν στον Γκένον Γένσεν, εκτελεστικό διευθυντή της ε, Συμμαχίας ε, την Γκένον Γένσεν του Health Environment Alliance. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που σας να, να μιλήσω πιο αργά με μεγάλη χαρά ε, δέχομαι, ε, δέχτηκα μάλλον την πρόσκληση ως ευκαιρία να μιλήσω ε, σε εσά σχετικά με το θέμα της υγείας συσχετιζόμενο με τις κλιματικές αλλαγές καθώς επίσης και τον οδικό χάρτη του 2050 που πραγματικά ελπίζομαι ότι θα λάβει υπόψη του την υγεία και την, τα ωφέλη και στο παρελθόν έχετε ασχοληθεί με ακραία φαινόμενα ε, περιβαλλοντικά ή του καιρού με ασθένειες οι οποίες σχετίζονται ε, με το κλίμα. Ε, είναι σημαντικό το θέμα της κλιματικής αλλαγής και ακόμα σημαντικότερα τα κέρδη που θα έχουμε εάν ξεπεράσουμε και το στόχο του 20% της κλιματικής αλλαγής. Η Συμμαχία της Υγείας και του Περιβάλλοντος έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο 65 και πλέον οργανισμών που εργάζονται έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη υγεία σε ένα υγιέστερο περιβάλλον. Ε, πρόκειται ε, για ομάδες ε, πολιτών, ασθενών, γυναικών, επαγγελματιών υγείας και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Το, από όταν ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το σύστημα ΧΙΛ, το 2007 μπορούμε να δώσουμε ε, στοιχεία που αφορούν ε, την ε, υγεία και να πούμε ότι η ε, ε, συνειδητοποίηση της ε, ιατρικής κοινότητας για το θέμα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκίνησε και την πρώτη της ημέρα υγείας για προστασία της υγείας σε σχέση με το περιβάλλον το 2007 και εκείνη την στιγμή το πρόγραμμα HIL κάλεσε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν περισσότερο φως στο θέμα αυτό. Προχωρώντας ακόμα περαιτέρω μπορούμε να πούμε πούμε ότι μπορούμε να έχουμε ακόμα περισσότερες ε, εξοικονομήσεις που να φτάσουν μάλιστα ε, σε πολύ υψηλά επίπεδα να ξεπεράσουμε τον στόχο του 20%. Ε, ποια είναι τα στοιχεία τα στα οποία έχουμε καταλήξει η νέα μας ε, μελέτη, την οποία έχουμε υποβάλει και στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, δείχνει με ε, ποσοστοποιημένο τρόπο τις, ε, τα ευεργετήματα και τα οικονομικά ωφέλη τα οποία ε, θα ε, απορρεύσουν από την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Καταδεικνύεται ότι με μείωση του 30% των εκπομπών οπωσδήποτε θα περιοριστούν οι μολυντές και επομένως θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Τα οικονομικά στοιχεία τα οποία ε, έχουμε ε, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ότι τα οικονομικά στοιχεία μπορεί να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο, ακόμα και σε σχέση με την έκθεση ΠΙΚ, ε, η οποία δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της ε, τα ωφέλη θα μπορούσαν να φτάσουν στα 30,5 δις ε, δηλαδή ε, που ισούνται με το 0,2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζω ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε παραπάνω από 52 δις εξοικονομήσεις για θέματα υγείας εάν προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα στόχο που θα ξεπεράσει τον σημερινό στόχο του 20%. Αυτή η νέα ανάλυση καλύπτει και το κόστος της αποφυγής θανάτου ή ε, ε, κάποιων ε, ασθενειών, όπως ας πούμε καλύπτει και το κόστος της μειωμένης δραστηριότητας λόγω προβλημάτων καρδιάς ή πνευμονικών προβλημάτων, το κόστος νοσοκομιακής περίθαλψης, το κόστος των επισκέψεων των, σε, γιατρούς ή το κόστος των φαρμάκων και προχωρούν ακόμα περισσότερο από τα στοιχεία που έδωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ίδια έκθεση αναφέρονται, ότι, ε, αναφέρονται λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία για 16 επιπλέον χώρες, ε, για το Βέλγιο, την Πολωνία, την Ουγγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, βεβαίως ε, το κέρδος για την υγεία θα είναι ακόμα μεγαλύτερο εάν αυξηθούν οι εξωτερικοί στόχοι. Και ε, το, τα υψηλότερα επίπεδα κέρδους του, των 30,5 δις αναέτος μέχρι το 2020 αναφυσούνται ε, με τα δύο τρίτα των εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το συνολικό κόστος εφαρμογής του στόχου του 30%. Ε, επιπλέον μπορούμε να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα εάν ξεκινήσουμε τη δράση μας τώρα. Ε, σύμφωνα και με τη μελέτη, εάν έχουμε περικοπή του 30% ε, του εγχώριου στόχου, τότε μπορούμε να φτάσουμε σε συνοφέλη για την υγεία που θα ξεπεράσουν το 250% σχετιζόμενο με το εάν θα ξεκινήσουμε τώρα τη δράση μας ή σε 5 χρόνια οι κυβερνήσεις ε, μπορούν ε, να περικόψουν τους προϋπολογισμούς ε, υγείας μέσω αποφυγής μελλοντικών ασθενειών και μελλοντικών ασθενών. Εάν ξεπεράσουν το στόχο του 20% σχετικά με την μείωση των εκπομπών, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μειώσουν σημαντικότατα το κόστος των αναπνευστικών ε, προβλημάτων ε, που βεβαίως ε, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο λαμβάνοντας υπόψη τον γυράσκοντα πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όμως όλα αυτά τα ωφέλη σε σχέση με την υγεία τα οποία ανέφερα, ανέφερα μέχρι τώρα αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου και το λέω αυτό γιατί τα συνοφέλη ε, ε, τα οποία, στα οποία θα μπορούμε να ε, καταλήξουμε εάν βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα ας πούμε μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερα. Ε, σε μια υγιή κοινωνία οι άνθρωποι βαδίζουν περισσότερο, κάνουν περισσότερο ποδήλατο ε, και επομένως ε, αποφεύγουν αρρώστιες όπως είναι η παχυσαρκία, ο διαβήτης, εγκυοκαρδιακές παθήσεις, ακόμα και κατάθλιψη θα θέλαμε να μεταφέρουμε τα αποτελέσματα, τα ευρήματα των μελετών μας ε, στο, στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε και αυτά με τη σειρά τους να τα μεταφέρουν στις εκλογικές τους ε, περιφέρειες. Ε, αυτή τη στιγμή η ιατρική κοινότητα αλλά και οι απλοί πολίτες στρέφουν το βλέμμα τους προς εσάς έτσι ώστε να οδηγήσετε σε μια ε, κοινωνία ε, με καλύτερη υγεία όπου και οι κλιματικές αλλαγές ε, θα οδηγούν σε ακόμα καλύτερη επίτευξη των οικονομικών στόχων και στόχων υγείας. Uh, uh, Ευχαριστώ που ήσασταν έτσι ήπια. Τελευταίος είναι ο Τζέισον Άντρισον επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κλιματικής και Ενεργειακής Πολιτικής στο ΒΒΕΦ και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευχαριστώ. Θα δω τι μπορώ να κάνω για τους διερμηνείς. Είναι ευχαρίστηση που έχω την ευκαιρία να μιλήσω εδώ πέρα σήμερα. Το ερώτημα που αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο είναι το εάν πρέπει να ζητήσει αύξηση του στόχου από το 20% στο 30% της Ευρώπης για να καταλήξει βεβαίως σε μια πολιτικά υπεύθυνη απάντηση πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής. Πρώτα απ' όλα, το εάν η περαιτέρω μίεση είναι αναγκαία για να αποφύγουμε την επικίνδυνη κλιματική αλλαγή. Δεύτερον, εάν χρειάζεται ένας στόχος για να επιτύχουμε περαιτέρω μειώσεις και τρίτον εάν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες υπέρ ή κατά ενός τέτοιου στόχου. Η πρώτη απάντηση είναι σαφής. Για να μην ξεπεράσουμε τους δύο βαθμούς, ε, το IPC όπως, είπε, όπως είπαμε μιλάει για μείωση 25 έως 40% και άρα εκεί πέρα το μερίδιο της Ευρώπης θα είναι γύρω στο 30% και με τα τωρινά δεδομένα θα ξεπράσουμε του τρει βαθμούς, κατά το οποίο θα είναι καταστροφικό η Ευρώπη. Δεν πρέπει να πώ. δεν παίζουμε πόκα εδώ πέρα. Μιλάμε για την επιβίωση του πλανήτη υπό τη μορφή που την ε, ξέρουμε. Η αλήθεια αυτή θα πρέπει να υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά μας. Το δεύτερο ερώτημα αφορά τον ρόλο των στόχων υπολογίζεται πως έχουμε επιτύχει 17,3% μειώσεις σε σχέση με το 1990 και να πω ό,τι φαίνεται πως μετά την οικονομική κρίση δεν θα επανέλθουμε στα προηγούμενα. Υπάρχει ε, βεβαίως ε, υπάρχουν 2,3 γιγατόνι σε άδειε ε, για συμμόρφωση, οπότε θα επιτύχουμε ούτως ή άλλως τον στόχο 20%, οπότε δεν χρειάζεται περαιτέρω ε, αυστηροποίηση του στόχου. Δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε άμεση και μισή κατεύθυνση για τη φιλοδοξία. Πρώτα απ' όλα το να κάνουμε πιο αυστηρό το στόχο είναι βασικό κίνητρο για το ε, σύστημα εμπορίας γιατί οι, δωρεάν άδειε έχουν δώσει έκτακτα κέρδη σε κάποιες βιομηχανίες ενώ ε, έχουμε έργα τα οποία δεν έχουν επιτύχει πραγματική μείωση των εκπομπών. Επιπλέον ε, θα μειωθεί και άλλο η τιμή του άνθρακα και αντί για το βασικό κίνητρο ε, εξυγχρονισμού θα καταλήξουμε σε μία υποσημείωση στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και άρα η αναθεωρημένη ε, βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να γίνει παραδείγματος χάρη δεσμευτική. Η αποτυχία των ε, εθελοντικών στόχων ή η τωρινή τάση να μην επιτυγχάνουμε τους μη δεσμευτικούς στόχους ε, μας δείχνει το τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν πραγματικοί στόχοι. Φτάνουμε στο τρίτο σημείο. Αν υπάρχουν άλλοι λόγοι υπέρ ή κατά ενό αυξημένου στόχου. Ακούσαμε, μα είπαν πω ε, το 30% κοστίζει πάρα πολύ. Η Ευρώπη είναι ήδη πρωτοπόρο. Η Ευρώπη δεν έχει πια καμιά σημασία στον κόσμο κτλ. Αυτά είναι αντιπερισπασμό. Γεγονό είναι πω ε, λίγα μέρη της ευρωπαϊκής οικονομίας επηρεάζονται στην ανταγωνιστικότητά της από την κλιματική πολιτική και προστατεύονται από την πολιτική αυτή και έχουν ε, από τις δωρεάν άδειες και οικονομικό όφελος. Όσον αφορά δε το μερίδιο της Ευρώπης είναι το εάν μιλάμε για ένα βάρος ή για ευκαιρία. Πολλές μελέτες ε, τονίζουν το πώς μπορούμε να επιτύχουμε μια νέα υφόρο οικονομία με ηγετικό ρόλο της Ευρώπης. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ έβγαλε μια έκθεση που λέγεται προς μια πράσινη οικονομία η οποία λέει πως θα οδηγηθούμε σε αυξημένες θέσεις εργασίας και θα μειωθούν βεβαίω οι κίνδυνοι του εάν κάνουμε τα ίδια με τώρα. Την περασμένη Δευτέρα το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ανάλογη έκθεση. Οπότε το μέλλον είναι αυτό το οποίο φτιάχνουμε. Πιο φιλόδοξος στόχος λοιπόν αποτελεί ένα βασικό κομμάτι ενός θετικού κύκλου που θα μας οδηγήσει σε μια οικονομία απομακρυσμένη από τον άνθρακα και θα οδηγηθούμε σε αύξηση του ΑΕΠ. Η διαδικασία αυτή δεν σημαίνει πως θα φύγουν οι βιομηχανίες από την Ευρώπη, είναι το νέο κύμα εκβιομηχάνησης και επενδύσεων. Στι αρχές αυτού του μήνα οι Barclays και η Accenture παρασίασαν νούμερα για το τι χρειάζεται να επενδυθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είπαν πως πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα στους επενδυτές το δίκτυο για την κλιματική δράση της Ευρώπης για το τσιμέντο, χαρτί και χάλιβα είπε πως οι τεχνολογίες του αύριο ήδη χρησιμοποιούνται. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι επενδύσεις και οι επενδύσεις αυτές θα έρθουν ακριβώς μέσω, τα, μέσα, των μέσων εκείνων από τους στόχους Ευρώπης. Βεβαίως αυτό δεν αρκεί από μόνο του αλλά είναι, είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη. Και βεβαίως, ενώ κάποιοι λένε πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να φύγει πολύ μπροστά από τους ανταγωνιστές της, τα στοιχεία πάνε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν για τον αντίκτυπο του ΑΕΠ, η Κομισιόν θα έπρεπε να πάει στο 30% για να ισοφαρίσει τις προσπάθειες άλλων οικονομιών και πάλι θα ήταν πίσω από Κίνα και Ινδία. Αν δείτε το επόμενο πενταετές κινέζικο σχέδιο, βλέπουμε πώς θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Σύμφωνα με την E3G, μιλάει για μια αύξηση δυναμικότητα 40% στις ΑΠΕ Κίνα. Μιλάμε δηλαδή για επενδύσεις τάξεως 20 πλάσιας από αυτήν της Ευρώπης. Το ίδιο και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. παίξει λοιπόν ένα ρόλο στην παγκόσμια σκηνή Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα και τα κίνητρα αυτά είναι ο στόχο του 30% στι εσωτερικέ μειώσει. Συνελώντη, Ιππίν. Το κοινοβούλιο σα θα έχει ω κίνητρο το φόβο ή την ευκαιρία. Θα υποκύψει στον εκφοβισμό ή θα επιδείξει αυτό το οποίο έδειξε τον περασμένο Νοέμβριο όταν κατέληξε στο 30% ή το Δεκέμβριο όταν ζήτησε δεσμευτικό στόχο μείωση. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Βόρεια Αφρική ε, δίνουν δύο σημαντικά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα πως είναι επικίνδυνη η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Αυξάνεται συνεχώς η ε, τιμή του πετρελαίου και άρα ήδη οι περσινές αναλύσεις είναι παροχημένες. Δεύτερον, κάτι το οποίο για μένα είναι μεγάλη έμπνευση. Οι απλοί άνθρωποι αντιστέκονται στα στρατεύματα πλησμένοι μόνο με πανό και αλλάζουν την ε, πορεία της ιστορίας και δεν κοιτάνε τις δυνατότητες ορμάνε προς το μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει λοιπόν να αποτρέψει αυτή την καταστροφή της κλιματικής αλλαγής και σας προτείνω να την αντιμετωπίσετε αυτή την πρόκληση κατά μέτωπον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε ο δεύτερος γύρος ε, μας έδωσε και άλλα επιχειρήματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Οπότε περνάμε τώρα στις ερωτήσεις. Περνάμε τον Καρλ Χάιντς Φλόρεντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, τον τελευταίο γύρο των παρεμβάσεων τότε η ευρωπαϊκή βιομηχανία μπορεί να αρχίσει να ανοίγει σαμπάνιες με το 30% γιατί θα έχει τελικά θετικά αποτελέσματα. Τουλάχιστον αυτό μας είπαν οι συνομιλητές μας. Και οι Γερμανοί επιστήμονες, οι οποίοι μίλησαν σήμερα όλοι αγγλικά παρόλα αυτά. Εμείς βεβαίως πρέπει να προσέχουμε γιατί πρέπει να επανεκλεγούμε και οι κύριοι αυτοί όχι. Αλλά η Κομισιόν ε, από ό,τι φαίνεται έχει απομακρυνθεί από το 30% και τώρα θα δούμε τι θα κάνει, θα απομακρυνθεί και το Κοινοβούλιο, τι θα προτείνει το Κοινοβούλιο. Για εμένα ε, με ενδιαφέρει περισσότερο η στόχη της αποτελεσματικότητας, αν θα πρέπει να είναι δεσμευτική ή όχι. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε γιατί όλοι γνωρίζουν στην Επιτροπή μας πως εγώ είμαι υπέρ της εφαρμογής των νόμων στα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο δεν γίνεται ούτε στον τομέα του κλίματος. Οπότε πώς το βλέπει αυτό ε, η συγγήτρια και, η, και η Κομισιόν, η οποία δυστυχώς βεβαίως τώρα πια δεν ε, μπορεί να απαντήσει. Ναι. Ε, μπορείτε να μιλάτε ό,τι γλώσσα θέλετε εδώ μέσα και, ισπανικά άμα θέλετε. Α, προσπαθήστε εσείς να επανεκλεγείτε με ισπανικά στη Γερμανία. Ε, ε, πρέπει να μιλήσω γερμανικά, καταλαβαίνετε. Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, Westlund. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω και εγώ σου ειδικά λοιπόν αφού είναι έτσι. Μία ερώτηση πρώτα απ' όλα για τον Άξελ Έγκερτ. Είπατε ξεκινώντας την παρέμβασή σας ότι εκπροσωπείτε ε, μία βιομηχανία η οποία θέλει να γίνει λιγότερο ενεργοβόρα ε, και η οποία θέλει να συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Ε, με ποιο τρόπο θα το κάνετε. Θέλετε να μας πείτε, μπορείτε να μας πείτε τι είναι άποψή σας σχετικά με αυτό που έλεγε ο κύριος Γκρουμπ, ο οποίος ε, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο άμεσης φορολόγησης ε, ε, των εισαγωγών σε περίπτωση διαρροής ή επανεισαγωγής των εξαχθέντων, του εξαχθέντος άνθρακος. Άλλη μια ερώτηση στην κυρία Γένσεν. Ε, από ό,τι κατάλαβα λέτε ότι οποιαδήποτε μείωση ε, του διοξιδίου του άνθρακος είναι καλή για την υγεία. Ε, όμως Ε, υπάρχουν ε, οι κινητήρες ε, αυτοί οι οποίοι όταν μπορεί να μειωθούν οι εκπομπές στο διοξείδιο του άνθρακος αλλά αυξάνονται οι εκπομπές άλλων μολυντών, άλλων ρήπων που είναι πολύ επικίνδυνοι για την υγεία. Επομένως τι μπορείτε να μας προτείνετε έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, τις καλύτερες επιπτώσεις για την υγεία. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τα πλεονεκτήματα του 30% στην υγεία και στις εργασίες. Είναι σημαντικό να δούμε και την κοινωνική πτυχή. Και εγώ, όπως ο κύριος Φλόρεντς, είμαι υπέρ της δεσμευτικής νομοθεσίας και θα ήθελα να θέσω το ερώτημα στους ειδικούς πρώτα απ' όλα ποια αποτελέσματα θα έχει η αυστηρή νομοθεσία στα κράτη-μέλη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μια νομική απέτηση για ανανεώσιμες φυγές ενέργειας και ένα ερώτημα ακόμα προς την Κομισιόν. Πόσο ε, δεσμευτική θα είναι η επίτευξη του 30% θα μπορούσε να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους εμπειρογνώμονες. Σε πολλά θα ήθελα να πω. Αλλά θα ήθελα ε, να ζητήσω το εκπρόσωπο της, ε, των βιομηχανιών Σιδήρου και Χάλιβα. Από όσο, από γνωρίζουμε για τον οδικό χάρτη, ε, γίνεται λόγος για μια αντιστάθμιση των, χωρών, των θέσεων εργασίας, συγγνώμη, αυτών που χάνονται δηλαδή και αυτών που θα ε, δημιουργηθούν. Ε, γίνεται λόγος για 2 εκατομμύρια θέσεων εργασίας, μέχρι και τα 6 εκατομμύρια φτάνουν. Θα ήθελα την άποψή του. να ρωτήσω και τον κύριο Άντερσον το εξής. Κατά την άποψή μου έχουμε δύο διαφορετικές στρατηγικές, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Από τη μία Ευρωπαϊκή Ένωση και από την την οι ε, υπόλοιπε χώρε. Εμεί έχουμε δεσμευτική στρατηγική, οι άλλοι έχουν τη στρατηγική ε, των, ε, της καινοτομίας, της έρευνας κτλ. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο δύο αντίθετες απόψεις σχετικά με την άλλη και η ηλική προσέγγιση. Εάν αφήσουμε όμως την βιομηχανία ελεύθερη, δεν πιστεύετε ότι θα υπάρχει μια απώλεια όσον αφορά την τεχνολογία. Ευχαριστώ. Μία σύντομη ερώτηση στον κύριο Έγκερτ. Ε, μας καταδείξατε το εσφαλμένο των μοντέλων της Επιτροπής. Ε, μήπως ε, μπορείτε όμως να μου πείτε κάτι παραπάνω σχετικά με την διαρροή άνθρακα ε, γιατί και σε σχέση με αυτά που είπε και ο κύριος Γκράμπ, ο οποίος φαίνεται ότι έχει την ίδια ε, αντίληψη όσον αφορά την διαρροή ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την κυρία Ντίξον. Έχετε πολλούς επενδυτές στον όμιλό σας ε, και ε, ξέρω ότι πέρσι βάλετε την ε, Κίνα στο, στην πρώτη θέση των επενδυτών με Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν σε σχέση με τα θέματα που συζητούμε σήμερα θα μπορούσατε να είστε λίγο πιο ασφαλείς όσον αφορά τις χώρες οι οποίες μπορεί να έχουν περισσότερα ωφέλη και τις άλλες. Ε, ε, αυτή την ερώτηση την κυρία Γένσεν. Ε, στον κύριο Άντερσον βεβαίως έχουμε και το πενταετές οικονομικό πρόγραμμα της Κίνας. Μπορείτε να μας πείτε κάτι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει, κάτι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πενταετές σχέδιο της Κίνας σε σχέση με το παγκόσμιο πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Αυτά. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση, κύριε Χασί. Ευχαριστώ. Οι δηλώσει του κυρίου Έγκερτ έρχονται σε μεγάλη αντίθεση με αυτά που ακούσαμε από τον καθηγητή Μάικελ Γκράμπ. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσει ο καθηγητής Γκράμπ ε, τα λεγόμενα του κυρίου Έγκερτ. Yeah. Ähm, äh, um, äh, είπατε πως εκπροσωπείτε προοδευτικούς ε, επιχειρηματίες. Ήταν εκεί πέρα, μου προξένησε εντύπωση, τράπεζες, ασφάλειες, Deutsche Telekom, είναι τομείς που δεν παράγουν τίποτα. Ε, δεν ε, ασχολούνται με πρώτες ύλε. Ε, είναι σε άλλους τομείς. Οπότε στις εκπροσώπους αυτούς υπάρχουν εταιρείες εκτός Ευρώπης. Και ποια είναι η σχέση μεταξύ των κλάδων που χρησιμοποιούν πρωτεσίλες και αυτών που δεν χρησιμοποιούν κατόπιν. Ο κ. Άντρισον είπε σύμφωνα με την εκτίμησή του οι πιστώσεις αυτές δεν οδήγησαν σε μείωση των εκπομπών μέχρι στιγμής. Δηλαδή το σύστημά μας δεν ε, έχει επιφέρει μείωση των εκπομπών. Μετά ο Dr. Turner είχε πει πριν πως και όμως αλλάζουν οι επενδυτικές συμπεριφορές όταν ε, σχεδιάζονται τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Λοιπόν, οπότε καταλήγουμε στις τελευταίες απαντήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τον Άξελ Έγκερ, 2 έως 3 λεπτά, νομίζω επαρκεί ο χρόνος. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτο ερώτημα από την κυρία Βέστλουντ για το τι προτείνουμε. Πρώτα απ' όλα, για να απαντήσω και σε κάποιες παρατηρήσεις του Leaders Group του πρίγκιπα της Ουαλίας. Οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας έχουν μειώσει ήδη κατά πολύ τις εκπομπές από το 1990 μέχρι το 2020 θα έχουμε μείωση πάνω από 40%. Είναι παραπάνω από αυτά που ζητάει το IPCC. Ποιος τα, τα έχει κάνει αυτά άλλος. Μάλλον θα είμαστε οι μόνοι που ανταγωνιζόμαστε και διεθνώς. Για το χάλιβα με Αυτό το οποίο είπε ο Τζέισον αφορούσε και το ερώτημα της κυρίας Βέσλουντ πως οι χαλιβουργίες έχουν ήδη νέες πειραματικές τεχνολογίες. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Η έκθεση του Climate Action Network δεν λέει κάτι τέτοιο. Είναι εκεί πέρα και το υποστηρίζουμε πως οι τεχνολογίες αυτές δεν θα είναι διαθέσιμες παρά μόνο το 2025 με 30 κάποιες ίσως νωρίτερα, αλλά με, μιλάμε για δέσμευση και αποθήκευση. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται υποδομή που πρέπει να μας τη δώσουν τα κράτη-μέλη. Και ξέρετε πως υπάρχουν τεράστια προβλήματα και επιπλέον αυτό πρέπει να συμφέρει κιόλα. Για τα μέτρα που προτείνουμε. Συγκεκριμένα πως θα πρέπει να υπάρχει σημαντική αύξηση και στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης στην πιλωτική φάση, φάση επίδειξης, αλλά και στο να μοιραστούμε την διαχείριση κινδύνου. Δηλαδή αν ε, επενδύουμε 500 εκατομμύρια σε ένα έργο και αποτυγχάνει, ποιος μοιράζεται μαζί μας τον κίνδυνο. Για τους στόχους χαλιβουργιών και άλλων κλάδων, θα ήθελα να ρωτήσω οποιονδήποτε εδώ μέσα, δώστε μας τεχνολογία. Εάν έχετε τεχνολογία, να δούμε και αν συμφέρει. Εάν συμφέρει και υπάρχει τεχνολογία, να την εφαρμόσουμε. Δώστε μας τεχνολογία όμως. Αυτό ήταν το, το ερώτημα. Ε, μετά υπήρχε ένα άλλο ερώτημα για εξαγωγικές επιστροφές, δασμούς. Ε, κάποια κράτη-μέλη μπορούν να διαφωνούν, αλλά τα περισσότερα από τα δικά μας μέλη λένε πως το μέσο αυτό δεν ε, θα εφαρμοστεί, θα μπλέξουμε με τις τρίτες χώρες. Θα είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε το, το όριο. Δηλαδή, εάν βάλουμε δασμούς ε, οι εξαγωγικές επιστροφές σε ένα τόνο χάλιβα, τι, τι κάνουμε με τα αμάξια. Στο κάθε αμάξι έχει 500 κιλά χάλιβα. Θα βάλετε και σε αυτό δασμούς. Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε. Δεν είμαστε, ως χαλιβουργία λέω τώρα, δεν είμαστε κατά των μέτρων ε, αντιστάθμισης στα σύνορα, αλλά μόνο εάν προσθεθούν με τις δωρεάν άδειες. Μετά υπήρξε ένα ερώτημα της κυρίας Γκαρντίνη για την απασχόληση. Βεβαίως αφενός θα ε, ε, Υπάρχουν ωφέλη, αφετέρου θα χάσουμε απασχόληση, αλλά κάποιοι λένε μιλάμε για ένα εκατομμύριο με έξι εκατομμύρια ε, Πού θα βρείτε όλους αυτούς τους εργαζόμενους ειδικευμένους. Ήδη σήμερα έχουμε προβλήματα να βρούμε αυτούς τους εργαζόμενους. Μετά ο κύριος Άικχαουτ για τη διαρροή άνθρακα. Πρέπει να είμαι πιο ακριβής. Ε, μιλάμε συγκεκριμένα για τα μοντέλα της Κομισιόν τα οποία χρησιμοποιούν τον λόγο 100% της τιμής. Αυτό δεν ισχύει για τομείς που κινδυνεύουν με διαρροή του άνθρακα. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ πέρα. Θα, θα, θα το, θα πέρναγα το κόστος και θα τελειώνει εκεί η υπόθεση. Μάλιστα, σε ευχαριστώ και, ζητώ συγγνώμη για το πόσο γρήγορα διάβασα την ομιλία μου. Πρώτα απ' όλα συμφωνούμε πως έχουν μειωθεί οι εκπομπές και καταβάλλονται προσπάθειες από τις βιομηχανίες ένταση ενέργειας και οπωσδήποτε τα δικά μας τα μέλη δεν θέλουν να να μπλέξουν ε, σε καυγά μαζί σας. Πολλά μέλη μας είναι βιομηχανίες ένταση ενεργής και έρχομαι σε αυτό το οποίο λέτε κύριε Πρόεδρε σε σχέση με τα μέλη εκείνα τα οποία βασίζονται σε πρώτες ύλε αντίθεση με τα άλλα. Κάποια από τα μέλη μας βασίζονται πάρα πολύ. Η σύμεξ, η ΣΕΛ, ορυκτά καύσιμα. Ζητάμε εμείς από αυτές τις εταιρείε να αλλάξουν πλήρως το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Η διαφορά είναι Πώ είναι διατεθειμένες να πάνε προ αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό νομίζω είναι το βασικό. Α μιλήσουμε τώρα και για τι εταιρείε που βασίζονται σε φυσικού πόρου και στην, και στην τιμή του χάλιβα, όπως είναι η Σαν Ρινό παραδείγματος χάρη. Αντιλαμβάνονται όλοι πως θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τη βιομηχανία, οπότε είναι διατεθειμένες να δουν τους κατάλληλους μηχανισμούς για να βοηθήσουν αυτές τις εταιρείες που έχουν τις περισσότερες δυσκολίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επανερχόμαστε σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Γκρουμπ και με το οποίο συμφωνώ. Χρειαζόμαστε μία λύση για τις βιομηχανίες εκείνες που θα πληγούν περισσότερο. Αλλά εξίσου δεν θα πρέπει να μειώσουμε το όραμά μας γιατί ε, μιλάμε μόνο για αυτές τις βιομηχανίες και να μην κοιτάμε άλλες εταιρείες που είναι διατεθειμένες να ανταποκριθούν στην πρόκληση και να λάβουν ρίσκα. Αυτά θα τα αναλάβουν τώρα όλοι οι κλάδοι. Σαφώς θα υπάρχει δυσκολία στις μεταφορές και πρέπει να δούμε που μπορεί να γίνει αυτό εξηλεκτρισμός και πάλι οι ε, θα προτείνουν λύσεις στον τομέα της ενέργειας όπου σαφώς κάποιοι από τους παραγωγούς ε, με τα καύσιμα πάνε σε άλλες πηγές και προμηθευτές. Επιπλέον πρέπει να δούμε τι είναι διατεθειμένα να κάνουν τα κράτη-μέλη και εδώ πέρα συμφωνώ με τον κύριο Φλόρεντς και πρέπει να δούμε και τη δεσμευτική νομοθεσία όσον αφορά την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αλλά και όσον αφορά τις συζητήσεις για τις ανανεώσιμες, πάντα ξέραμε πως τα εθελοντικά μέτρα δεν λειτουργήσαν και άρα είναι πιο αποτελεσματική η υποχρεωτική δεσμευτική νομοθεσία για να οδηγηθούμε σε αλλαγή και επενδύσεις. Όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Έκχαρτ για το ότι οι Κινέζοι είναι οι πρώτε επενδύσεις, ναι, απολύτως σωστό. Αυτό δεν έχει απλά αλλάξει την επενδυτική αγορά, δεν έχουν απλά οι επενδυτές δει την Κίνα ως ε, ένα μέρος όπου θα γίνουν οι επενδυτικές αποφάσεις, αλλά με το πενταετές σχέδιο και με την ίση δημόσια χρηματοδότηση, ο ιδιωτικό τομέα θεωρεί την Κίνα την αγορά χαμηλού άνθρακα, όχι την Ευρώπη. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε ηγετικό ρόλο. Και όπω έχουν πει πολλοί από εμά, πρέπει να δούμε ισχυρού στόχου μαζί με ισχυρό σύστημα εμπορία και έτσι να ανέβει και η τιμή του άνθρακα και να έχουμε κίνητρα προς σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση ήταν σχετικά με αυτό που είπα εγώ ότι ό,τι είναι καλό για το κλίμα είναι καλό και για την υγεία. Εντάξει, δεν είναι 100%. Αυτό όμως που προσπαθούσα να πω είναι ότι πολλές δράσεις που πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να μειώσουμε τις εκπομπές είναι πράγματα από τα οποία θα αποφεληθεί και η υγεία. Θέλουμε να είμαστε πιο αποδοτικοί όσον αφορά την ενέργεια και συγχρόνως πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τέτοιων μέτρων στην υγεία των ανθρώπων. Μήπως υπάρχουν και ασθένειες. Άρα υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα. Προσπαθούμε πάντως να καταδείξουμε εδώ ότι λέμε ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές για να προστατεύσουμε τον πλανήτη, αλλά όχι μόνο, γιατί έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε και την υγεία του κόσμου και να του προσφέρουμε ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο θα χρησιμοποιεί λιγότερα αυτοκίνητα, θα έχει περισσότερους πράσινους χώρους στην πόλη του κλπ. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε ωφέλη και για την υγεία. Για την ερώτηση της κυρίας Βέσλιν τώρα, για το ποιο, ποιοι τομείς καταστρέφουν περισσότερο την υγεία. Η έκθεση που δεν κοίταξε επιτροπή, και εντάξει δεν είμαι εδώ εμπειρογνώμων, δεν θέλω να σχολιάσω, θα τις τα πω μετά της κυρίας Βέσλιν. Το τελευταίο ήταν ποιες χώρες θα υποφεληθούν περισσότερο αν πάμε στο 30%. Εδώ η έκθεση δείχνει ότι η Γερμανία, η Πολωνία και η Γαλλία και η Ιταλία είναι από εκείνους που θα υποφεληθούν περισσότερο. Και αυτό είτε γιατί έχουν μεγαλύτερο πληθυσμό ή γιατί και οι χώρες που βρίσκονται γύρω από αυτές θα υποφεληθούν από αυτό το υψηλότερο ποσοστό. Πάντα από την έκθεση φάνηκε ότι χώρες όπως είναι το Λουξεμβούργο, που έχει μικρό πληθυσμό, θα υποφεληθεί επίσης. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ο κύριος Άντερσον. Ρωτήσατε κατά πόσο το σύστημα εμπορίας οδηγεί σε μείωση των εκπομπών ή όχι. Είναι ένα περίπλοκο θέμα. Είναι δύσκολο να κάνουμε διάκριση και να πούμε πού οφείλεται αυτή η μείωση. Σίγουρα υπάρχει μια σωστή τάση. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα βοηθάει σε τέτοιο βαθμό που να αξίζει να του δώσουμε ένα καλό βαθμό. Να πούμε δηλαδή ότι ναι βοηθάει. 40% Μπορεί βέβαια ένα ποσοστό να οδηγεί σε αύξηση των εκπομπών αλλού. Οπότε είναι δύσκολο να πούμε ακριβώ ποιο είναι το ποσοστό της μείωσης που οφείλεται στο σύστημα. Ορισμένοι λένε ότι μόνο το 2017 μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά έχουμε μειώσεις. Ότι οι μειώσεις που παρατηρούνται σήμερα δεν είναι εξαιτίας ε, του συστήματος, αλλά εξαιτίας μιας ε, πολιτικής που ακολουθείτε. Το δεύτερο που με ρωτήσατε έχει να κάνει με την ε, φύση των μειώσεων στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες χώρες του κόσμου. Οι δεσμευτικοί στόχοι της Ευρώπης αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχει στη διαθέσή της η Ευρώπη και από το οποίο εμπνέονται κι άλλοι, έμεσα ή άμεσα. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση ίσως, αλλά σίγουρα η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει και στην έρευνα και να μην βάζει μόνο στόχους. Μια μελέτη δείχνει της PwC ότι χρειάζεστε ή έρευνα ή το αντίστοιχο σε στόχους. Εμείς λέμε ότι χρειαζόμαστε και τα δύο, και έρευνα και στόχους. Διαπίστωσαν πάντως ότι το πιο σημαντικό δεν ήταν η έρευνα και η ανάπτυξη, αλλά στόχοι στην αγορά που οδηγούν σε χρήση νέας τεχνολογίας από την αγορά. Κατά πόση τεχνολογία, στο χάλιβα, στο χαρτί κτλ πρέπει να περιμένουμε το 2025-2030, ε, δεν θα εμφανιστούν ξαφνικά διαθαύματα στην αγορά. Προηγουμένως χρειάζεται να υπάρχει μια τάση, έρευνα για να φτάσει στην εμπορεύσιμη τεχνολογία. Άρα από τώρα μέχρι το 2020 και με το 2030 ε, δεν βλέπω να υπάρχουν αυτές τις τεχνολογίες. Τα περιτιμών τα ξέραμε. Τέλος για τις διαπραγματεύσεις σε διεθνές επίπεδο με την Κίνα λοιπά Στο Κανκούρ για πρώτη φορά είδαμε να λαμβάνεται απόφαση από τα Ηνωμένα Έθνη. Πραγματικά. Είναι ένα βήμα που δεν φτάνει. Που δεν είναι το κατάλληλο. Γιατί υπάρχει τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις προτάσεις που γίνονται και στα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε για τους δύο βαθμούς. Χρειάζεται οικοδόμηση εμπιστοσύνης, εμβάθυνση στους στόχους. Υπάρχει η Κίνα, θα υπάρχουν και άλλες χώρες σαν την Κίνα, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρχουν η Ευρώπη και άλλες χώρες σαν την Ευρώπη με υψηλούς και φιλόδοξους στόχους. Οπότε στην επόμενη συνάντηση να μετρήσουν περισσότερο. Ευχαριστούμε. Και τέλος. Ναι, μου ζητήσατε να αναφερθώ στις διαφορές στο modeling. Λέω Σκραμπ. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση από εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρόλο που τα αποτελέσματα είναι λίγο πολύ τα ίδια. Δεν ξέρω γιατί υπάρχουν ό,τι διαφορές υπάρχουν, αλλά δεν είναι ουσιαστικές. Γιατί το modeling είναι για το τι θα γινόταν αν υπήρχε πληστηριασμός και δεν υπήρχαν δωρεάν δικαιώματα. Η πραγματικότητα είναι ότι κάνουμε πράγματα, δωρεάν δικαιώματα, ναι, εγώ δεν ξέρω αν συμπεριλαμβάνει στα νούμερά του ο κύριος Έγκαρτ και τα δωρεάν δικαιώματα. Πάντως, οι διάφορες βιομηχανίες πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για την μείωση χρήσης άνθρακα. Οι διορθώσεις είναι ένα πράγμα που πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο είναι να μην πρόκειται μόνο για τις πρώτες ύλε, αλλά και για παράγωγα. Και εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Αν πούμε ότι κάτι πρέπει να εφαρμοστεί παντού και στα πάντα, είναι καλύτερη συνταγή για να μην γίνει τίποτα. Και εδώ περί αυτού πρόκειται. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με μία κατηγορία προϊόντων, αυτά που εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα και σιγά σιγά να προχωρήσουμε. Τα ελεύθερα δικαιώματα δεν μπορείτε να ζητήσετε στα σύνορα αντιστάθμισμα. Υπάρχει το border leveling. Μέτρα τα οποία είναι απόλυτα συμβατά με τον ΠΟΕ. Και τα έχουμε συζητήσει με τον ΠΟΕ. Ο συνδυασμός των ε, πληστηριασμός με το border leveling είναι κάτι θεμητό. Και έτσι μπορούμε να πάμε στο 30% σίγουρα για το τσιμέντο, ίσως και για το χάλιβα, με αύξηση των εσόδων κατά 100 δις. Σίγουρα χρειάζονται και επενδύσεις στο χάλιβα σε συνδυασμό με όλα τα προηγούμενα. Ο Μπας πέρασε και η ώρα. Και σας δίνουμε και δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ για τα δύο λεπτά, ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα τώρα να πω τι θα κάνουμε μετά. Ήταν πάρα πολύ καλό που είχαμε όλες αυτές τις πληροφορίες και ευχαριστούμε όλους ε, για τα όσα μας είπαν, γιατί ακούσαμε και ε, την άποψη των επιστημόνων και την άποψη των ε, ΜΚΟ και την άποψη της βιομηχανίας και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τις απόψεις αυτές έτσι ώστε να έχουμε μια καλή σχέση με όλους τους ενδιαφερόμενους σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως σημαντικό είναι και η πληροφόρηση που θα έχουμε σε επίπεδο κρατών μελών ε, γιατί οι διαφορές θα πρέπει να αντισταθμιστούν μέσω ας πούμε της πολιτικής ε, σύνοχης. Ε, ακούσαμε τον κύριο Έγκερτ να εκφράζει ανησυχίες και επομένως θα πρέπει να βρούμε ένα σωστό βαθμό έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε πολιτικές push and pull. Θα ήθελα όμως να σα αφήσει επί του ε, εξής, ότι ε, ο συντονισμός ε, ε, των ελευθέρων ε, ποσοτήτων και το, της αντιστάθμισης στα σύνορα δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή θεωρούμε το Η κυρία Τζόρνταν και εγώ κάνουμε, κάνουμε, Τζορντάνα και εγώ κάνουμε δύο διαφορετικά δύο διαφορετικές εκθέσεις βλέπουμε το ίδιο θέμα από δύο διαφορετικές πλευρές. Στις 17 ε, σήμερα ακούσαμε τα θέματα πλευράς περιβαλλοντικής. 17 Μαρτίου θα έχουμε και την Επιτροπή Ήτρε που θα έχει τη δικιά της ε, ακρόαση. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να ετοιμαστούμε πριν από το τελικό ε, συμβούλιο που και η εκπρόσωπος της Ουγγρικής Προεδρίας μας είπε ότι θα είναι σημαντική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, ευχαριστώ λοιπόν τους 7 εμπειρογνώμονες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι τελευταίες μισή ώρες. Είχαμε πολύ υλικό λοιπόν για τις εκθέσεις μας και τις πολιτικές αποφάσεις. Εμένα μου φαίνεται πως το 20% είναι ένα σενάριο business as usual και η Ευρώπη μέχρι το 2020 μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα και θα είναι θα τα καταφέρει καλύτερα και θα πρέπει να ακολουθήσουμε φιλόδοξη γραμμή στο Κοινοβούλιο. Έως ε, θα πρέπει να προσέξουμε όσον αφορά τα μέσα, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Γιατί η έννοια του 2020 είναι, ξέρετε, smart, intelligent and sustainable growth. Έξυπνη, έφυης ε, και αηφόρος ανάπτυξη. Ακούσαμε τα επιχειρήματα και είμαι σίγουρος πως η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας θα κινηθούν σε μια γραμμή που θα καταλήξει σε πλειοψηφία ε, στην Ολομέλεια για να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι με τα 27 κρατημέλη μετά και την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν, ευχαριστώ τους ειδικούς, ευχαριστώ τους βουλευτές και όλους όσους άκουσαν για τη συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας.